We are just checking whether the Commission is here for the first agenda point and they are, they are here. Then uh, let's start. Ήρθε η Κομισιόν αγαπητοί συνάδελφοι, οπότε μπορούμε και εμείς να αρχίσουμε γιατί έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Αρχίζουμε με την έγκρισή της. Η έκθεση για την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον αναβάλλεται. Η έκθεση Κύρκοπ όμως για τα προσωπικά στοιχεία των επιβατών. 11.30 με 12.30 θα συζητηθεί σήμερα. Ο Έλληνας Υπουργό για την Προστασία του Πολίτη κύριος Χρυσοχοίδης θα προσέλθει το απόγευμα για να μας μιλήσει για την κατάσταση στην Ελλάδα ως προς τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. 3 με 4.30. 3 με 4 και η έκθεση της Europol θα παρουσιαστεί επίσης σήμερα μετά την ψηφοφορία 5.30 με 6.30. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται με το σχέδιο ημερήσιας διάταξη και γίνεται ημερήσια διάταξη. Ε, υπάρχουν και τρεις ανακοινώσεις. Οι συντονιστές συνέστησαν στην προηγούμενη του συνεδρίαση η κυρία Μακοβέη να είναι η συγγήτρια για την κατάσχεση εσόδων από το έγκλημα και ο κύριος Δρούτσας εισηγητής για την, προστασία, την οδηγία της προστασίας των δεδομένων μετά από πολλή συζήτηση. Αν δεν έχετε αντίρρηση εγκρίνουμε τις συστάσεις αυτές των συντονιστών. Είπαμε ότι θα ψηφίσουμε από τις 4 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Να μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Και τελευταία ανακοίνωση. Στην προηγούμενη Ολομέλεια ανακοινώθηκε ότι 12 παρατηρητές από την Κροατία θα προσέρχονταν και μία από αυτές η κυρία Ίγκριντ Αντιτσέβιτς Μάρινοβιτς είναι εκείνη που θα έρθει εδώ στη συνεδρίασή μας, δεν ξέρω αν έχει έρθει ήδη, όχι ακόμα, αλλά νομίζω στο δρόμο θα είναι. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το σημείο 3 προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό. Η συγγήτρια κυρία Εδίθ Μπάουερ. Υπάρχει και πρόσωπος της Κομισιόν. Θα αρχίσουμε με την παρουσίαση της Κομισιόν και μετά θα μιλήσει η κυρία Μπάουερ. Ορίστε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω και εγώ γιατί πρέπει να φύγω μετά. Εντάξει. Λοιπόν, η παρουσίαση της Κομισιόνου. που είναι Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό. Η σημασία του θέματος αυτό έχει γίνει προφανή στις τελευταίες κρίσεις όπως στη Συρία. Στη Λιβύη 6.000 πολίτες της Ένωσης ζούσαν όταν ξέσπασε η κρίση, αλλά υπάρχουν και πιο κανονικές καταστάσεις όπως η απώλεια διαβατηρίου. Οι πολίτες της Ένωσης που διαβιούν σε τρίτες χώρες όπου δεν υπάρχει κάποια ένωσια, όπου δεν υπάρχει προξενείο ή πρεσβεία της χώρας τους έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν σε προξενεία ή πρεσβείες άλλων ενωσιακών χωρών. Αυτό το προβλέπουν και οι συνθήκες και είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρει η χάρτα. Το δικαίωμα όμως αυτό έπρεπε να υλοποιηθεί πληρέστερα. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας προτείναμε αυτή την οδηγία η οποία ανταποκρίνεται και σε εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενδυνάμωση της προξενικής προστασίας μετά την θέση ενισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω λιγάκι το περιεχόμενό της. Δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για την προστασία από τις προξενικές αρχές και αποσαφηνίζει τα κύρια θέματα ώστε να μπορούν οι προξενικές αρχές και οι πολίτες να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, παραδείγματο χάρη. Ότι μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες μιας ενωσιακής χώρας να απευθυνθούν σε προξενείο άλλης και μάλιστα για κατεπήγοντα θέματα ταξιδίου κτλ. χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα όπου θα ίσως είναι η πρεσβεία και το προξενείο τους. Αυτό ισχύει ας πούμε για την Κίνα. Και είναι υποχρεωμένες οι προξενικές αρχές να τους προστατεύσουν σαν να ήταν οι πολίτες της δικής τους χώρας. Σε καταστάσεις κρίσεως προβλέπουμε να συγχρηματοδοτούνται οι εκενώσεις, οι μεταφορές πολιτών από ένα συγκεκριμένο ταμείο εν μία από τις χώρες μέλη που έχει προξενείο την ε, ενδιαφερόμενη χώρα θα αναλαμβάνει πάντοτε το συντονισμό. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα συνεννοούνται τακτικά για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια λογικότερη χρήση των πόρων που διαθέτουμε τέλος διευκολύνουμε και τις αποζημιώσεις, αποκινούμε όλα τα τη μελη Η διαδικασία αυτή αποζημιώσεων έχει σημαντικά απλοποιηθεί και βελτιώνει έτσι και τη συνεργασία μαζί με τις εξοικονομήσεις. Γενικά είναι θέμα η οδηγία αυτή ενωσιακής αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας και ελπίζουμε η Επιτροπή ΕΛΕΦ να μπορεί να την στηρίξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Τώρα το λόγο έχει η Εδίθ Μπάουερ. Πάρτε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ακόμα ένα βήμα έτσι ώστε να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών και νομίζω ότι θα αποτελούσε ε, μια καλή υλοποίηση του άρθρου 23 της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς επίσης ε, και την υλοποίηση ενός από τους στόχους του προγράμματος της Στοκχόλμης. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν σε αυτό το πεδίο ε, ε, ισχύουν διάφορες συνθήκες και αποφάσεις. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποια πρακτικά ε, σημεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να αποσαφινιστούν σε σχέση <clears throat> με αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης για το ζήτημα που μας απασχολεί. Για παράδειγμα, απαραίτητο είναι να αποσαφινιστεί ποια είναι η, απαραίτητη, η προστιθέμενη αξία σε σχέση με την 553 του 93. Επίσης να αποσαφινιστεί ποια είναι η σχέση ε, με τα άρθρα 36-37 της Συνθήκης της Βιέννης όσον αφορά τα μέλη οικογενειών από ε, υπηκών τρίτων χωρών όσον αφορά τις ε, χρηματοδοτικές διαδικασίες ε, και ε, το μοίρασμα του άχθους. Επίσης, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν οι διάφορες πρακτικές των κρατών μελών διότι η προξενική αρρωγή σε μερικές χώρες είναι δωρεάν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι. Ε, κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχουν κάποια πρακτικά σημεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να αποσαφινιστούν στη διάρκεια της ε, συζήτησης. Και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συμφωνία κυρίως μεταξύ των μεγάλων κρατών μελών διότι για να σας μιλήσω ειλικρινά, το το μεγαλύτερο άχθος ε, θα αφορά αυτές τις μεγάλες χώρες. Να υπενθυμίσω ότι τρεις χώρες στον κόσμο είναι τέτοιες που έχουν εκπροσώπους τους σε όλες τις χώρες μέλη και επομένως ε, αυτοί θα στηρίξουν, θα, θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος. Είναι σαφές λοιπόν ότι ε, η διαδικασία αυτή θα αποβεί ε, προς όφελος των μικροτέρων χωρών αλλά το βάρος θα το σηκώσουν οι μεγαλύτερες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές εάν και εφόσον θέλουν να σχολιάσουν ή να υποβάλουν ερωτήσεις. Λουί Μισελ, ο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την παρουσίαση αυτής της οδηγίας, η οποία όντως είναι πολύ σημαντική για τους υπηκόους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν εκτός των συνόρων αυτής. Είναι σημαντικό επίσης ε, να υπάρξει ε, ε, δυνατότητα πρόσβασης στην προξενική αρρωγή για υπηκόους πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων η χώρα δεν εκπροσωπείται προξενικά. Όμως, οι διατάξεις της απόφασης 95 593 ε, ε, ε, δεν, δεν ασχολείται παρά μονάχα με μερικές όψεις της προβληματικής αυτής και επομένως θα πρέπει να αντικατασταθεί. Κάθε κρίση, οποιασδήποτε φύσης κι αν είναι αυτή, οπωσδήποτε δημιουργεί ανάγκες προξενικής αρρωγής. Το τσουνάμι ας πούμε στο Ισραήλ, το, στον Λίβανο, οι σεισμοί τρομεροί της Αιτής και της χείλη, καθώς επίσης ε, και το πρόβλημα που προκλήθηκε μετά από την έκθεση του ηφαιστείου στην Ισλανδία, καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μοίρασμα του βάρου μεταξύ των κρατών μελών. Ε, η ε, συγγνώμη, ο κανονισμός αυτός ε, δίνει απάντηση σε κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαβιούν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και υπάρχουν επίσης διατάξεις που αφορούν την βελτίωση της πρόσβασης στην προξενική αρρωγή υπηκών τρίτων χωρών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Βεβαίως καλύπτονται κυρίως τα προβλήματα των υπηκών των χωρών μελών που ζουν σε περίοδους σε και σε περιοχές κρίσης ε, χωρίς να έχουν προξενική αντιπροσώπευση της χώρας τους. Ε, παραμένουν επίση και κάποιες φαίες ζώνες. Ε, αναφέρεται σαφώς ότι οι πρεσβείες και τα προξενία βοηθούν του τους εκπροσώπους, τους πολίτες μάλλον μη εκπροσωπούμενων χωρών σαν να ήταν οι πολίτες των χωρών που εκπροσωπούνται. Υπάρχει τρόπος μέτρησης ή εργαλείο μηχανισμός μέτρησης ε, αυτής ε, της ε, πρότασης. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ότι δεν θα υπάρξει προτεραιότητα από τις προξενικές αρχές προς τους πολίτες της ίδιας της χώρας που εκπροσωπείται σε σχέση με τους πολίτες των χωρών που δεν εκπροσωπούνται προξενικά. Επίσης ποιος τελικά θα αναλάβει το μεγαλύτερο κόστος αυτής της αρρωγής θα πρέπει να υλοποιηθεί η οδηγία αυτή βάσει και των ε, ε, όσων αναφέρονται στο άρθρο 23 της Συνθήκης Λειτουργίας ε, να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση ακόμα και όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ας πούμε δεν αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ ομοφύλων. Συγγνώμη. επομένως τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση αν δηλαδή παρουσιαστεί μια ομόφυλη οικογένεια και, να και ζητήσει την προξενική αρρωγή. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ ελπίζω ότι πριν φύγετε θα μπορέσετε να λάβετε κάποιες αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. And, Η uh, ε, κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και την Επιτροπή την Κομισιόν που προσήλθε για να μας, πει την παρουσίαση, να μας κάνει την παρουσίαση της. Βέβαια, μια, μια οδηγία σαν και αυτήν είναι απαραίτητη ιδιαίτερα εν ώψη των τελευταίων γεγονότων που ανέφεραν και η Δίθ Μπάουρ και ο κύριος Μισελ. Συμφωνώ βέβαια με την πρόταση και με το οικονομικό της τμήμα, χρηματοδοτικό, και ρωτώ την Κομισιόν το εξής. Ξέρουμε ότι σε μερικές χώρες μέλη δεν υπάρχουν προξενία και αντιμετωπίζουν εκεί προβλήματα και αυτές θα ωφεληθούν ιδιαίτερα, αλλά ίσως χρειάζεται να αναφερθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για εκείνες. Επίσης για το... We have also... Επίσης για το εύρος εφαρμογής της οδηγίας, ποιους ακριβώς θα καλύπτει. Μιλήσατε για οικογένειες. Τα είπε και ο κύριος Μισελ, αλλά και αυτοί που καλύπτονται από τον κανονισμό 539 και εκείνους που έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης κόμμα υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που δεν καλύπτεται εδώ, δεν αναφέρεται. Οι πρόσφυγες οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία εθνικότητα που έχουν ή δεν έχουν διαβατήριο κάποιας χώρας μέλους που έχουν μάλλον διαβατήριο κάποιας χώρας μέλους ε, και οι Λετονοί και οι Εσθονοί έχουν τέτοιο πρόβλημα οι κάτοικοι της Λετονίας και της Εσθονίας πάνω από 15% εκεί δεν έχουν το εθνικό διαβατήριο. Μήπως υπήρξε κάποια παρεξήγηση λοιπόν, μήπως η Κομισιόν έχει κάποιο λόγο που δεν συμπεριέλαβε αυτούς τους ανθρώπους στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα για το πεδίο εφαρμογής. Ο κύριος Μπρόγκς. Τη διάβασα την έκθεση και είμαι υπέρ. υπέρ. Ελπίζω να μην σας σοκάρει αυτό με βάση τη φήμη που έχω δημιουργήσει, αλλά δεν νομίζω ότι η έννοια της ενωσιακής ηθαγένειας έχει πολύ μεγάλο παρελθόν. Σίγουρα όχι πριν τη συνθήκη της Μαστρίχτης. Η Σουηδία, η Νορβηγία και χώρες σαν αυτές που δεν είναι και χώρες που δεν είναι στην Ένωση όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφάρμοζαν ήδη αυτά τα μέτρα να προστατεύουν πολίτες χωρών που δεν είχαν προξενικές αρχές Ελπίζω μάλιστα οι πρεσβείες να βοηθούν γενικά τον κόσμο χωρίς να του ζητάνε το διαβατήριό του. Υπάρχει όμως και ένας κίνδυνος. Αν αρχίσουμε να μιλάμε και για πρόσφυγες κλπ, τότε οι πρεσβείες μπορεί να έχουν αντιρρήσεις να βοηθήσουν και τέτοιους ανθρώπους. Ευχαριστώ, δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο βλέπω. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην Κομισιόν, η σκιώδη Στάνια Φαγιάν μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός της. Υποστηρίζει γενικά τους στόχους της οδηγίας γιατί απλοποιεί τα πράγματα και τις διαδικασίες και πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών που μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ηθαγενείας και συνείδησης. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν διευρυμένο δίκτυο προξενικών αρχών στο εξωτερικό, ιδίως οι μικρότερες. δέχεται και την διάταξη που δίνει το δικαίωμα στα μέλη των οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ηθαγένεια τρίτης χώρας σε προξενική προστασία και θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη κάποια βελτίωση εδώ. Το είπαν και άλλοι. Δηλαδή, το κράτος που θα αναλαμβάνει το συντονισμό της αντιμετώπισης κρίσεων σε κάποια τρίτη χώρα, εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις και λέει ότι η Επιτροπή ΕΛΕΦ πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις συστάσεις που, θα κάνει το κοινο... που έχει κάνει το Κοινοβούλιο από το 2007 σε μία πράσινη βίβλο του για να υπάρξει πραγματικά εναρμονισμένη εφαρμογή της προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών στο εξωτερικό. Όπως σας είπα και πριν το 2007 το είχε ζητήσει ήδη το Κοινοβούλιο. Σε ψήφισμα λέει τώρα η ομιλήτρια, πριν ήταν πράσινη βίβλος. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντανιέλ Βόλ τώρα να απαντήσει ίσως μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν και μετά η συγγήτρια. Ευχαριστώ και για τα θετικά σχόλια που υπήρξαν μέχρι στιγμής για το οποίο είμαστε φυσικά ευγνώμονες. Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε Εάν ε, μπορούν να αναμειχθούν τα δικαστήρια, όπως λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ε, τον ε, Μάρτιο, το άρθρο 3 εφαρμόζεται ήδη. Ένας πολίτης λοιπόν που θα αιτείται προξενική βοήθεια θα μπορούσε να διωχθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε ωστόσο να υπάρχει επαρκής δυνατότητα εκένωσης να μπορούν να αποχωρήσουν όλοι οι πολίτες. Άρα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο κενό για τον σεξουαλικό προσανατολισμό των μελών της οικογένειας. Η σκέψη 9 της οδηγίας που αναφέρεται στην 2004-48 ε, οδηγία όπου λέγεται ότι για τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να εμπνεόμαστε από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας όπου αναφερόμαστε σε οικογενειακές σχέσεις ε, ιδίου φύλου. Για την ε, κατανομή του οικονομικού κόστους και άλλων βαρών προβλέπεται να υπάρχουν επιτόπου ρυθμίσεις και ιδιαίτερα διμερεί μεταξύ κρατών μελών, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη επιτόπου να μπορούν να κατανέμουν το βάρος αρρωγή. Ένα κράτο μέλος, για παράδειγμα, μπορεί να ασχοληθεί με κάποιε εθνικότητες, άλλο με κάποιες άλλε. Είναι δυνατό λοιπόν αυτό, αλλά και σκόπιμο εφόσον δεν ε, εμποδίζει την αποτελεσματική ε, προστασία και εφόσον είναι διαφανείς αυτές οι ρυθμίσεις. Και μπορούμε να συζητήσουμε αν επαρκούν αυτά ή όχι. Όσον αφορά το εύρος εφαρμογής ε, για τα μέλη της οικογένειας, εάν συμπεριλαμβάνονται οι απάτριδες, οι πρόσφυγες και άλλες παρόμοιες κατηγορίες. Πρέπει να σεβαστούμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο που βασίζεται στο άρθρο 23 για την ηθαγένεια. Ηθαγένεια Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα και στο ποια μπορεί να είναι τα μέλη της οικογένειας. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα τα σκόπουμε να συμπεριλάβουμε και ευρύτερο ε, τμήμα των ε, συνδεωμένων με τα, τους πολίτες της Ένωσης. Ελπίζω να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο μαζί μας. Ποιο θα είναι το κράτος που θα έχει τον πρώτο ρόλο, το ηγετικό κράτος. Νομίζω ότι είναι ήδη αρκετά λεπτομερείς ε, οι αναφορές που κάνουμε για το θέμα αυτό. Αν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση, να ακούσουμε περαιτέρω ε, προτάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει ε, αυτά που νομίζουμε ότι είναι ρεαλιστικά και αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν λοιπόν στην πράξη. Για την τελευταία ερώτηση για την εναρμόνιση θεμελιωδών δικαιωμάτων να επαναλάβω ότι το άρθρο 23 μιλάει για, ε, για το δικαίωμα μη διακρίσεων. Δηλαδή, οι πολίτες πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ε, ισότιμα με τους πολίτες του κράτους. Άρα δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω εναρμόνισης, εφόσον είμαστε υπέρ της ε, ισότιμης μεταχείρισης και της, ε, των μη διακρίσεων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Έντιτ Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Τονίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη πολλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επί της αρχής κάποιο πρόβλημα αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η οδηγία. Διότι τα διάφορα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά τις διάφορες διατάξεις, διότι έχουν διαφορετικές δομές και νοοτροπία. Για παράδειγμα, πώς θα προλάβουμε καταστάσεις όπου τα προξενία στα οποία θα στραφούν οι πολίτες Ε, μπορεί να πάρουν χρήματα από τους πολίτες άλλων κρατών ενώ δεν παίρνουν από τους δικούς τους πολίτες. Να δούμε τις ε, διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης που καθορίζει ότι τα μέλη των οικογενειών πολιτών τρίτων χωρών καλύπτονται. Κάποιοι μπορεί να έχουν συλληφθεί ή σε καταστάσεις ε, κρίσης. Θα προκύψουν πρακτικά ζητήματα και η μεγαλύτερη δυσχέρεια θα είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, συνεπής εφαρμογή των νόμων και ε, εναρμόνιση και συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων και άρθρων. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον. Αυτά θα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Και όπως είπα, οι αρχές είναι ορθές. Αλλά το πώς θα ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε κρίσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Υπάρχουν κάποιες νέες ε, αρχές, ορισμένοι νέοι όροι. Ποιο θα είναι το ηγετικό κράτος. Θα παίξει σημαντικό ρόλο σε περίπτωση κρίσης. Άρα το θέμα είναι και βεβαίω τα καθημερινά προβλήματα, τα πρακτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα διασφαλίσουμε αποτελεσματική προστασία σε περιπτώσεις καταστάσεων κρίσης. Προσβλέπω λοιπόν σε καρποφόρα και επικοδομητική συνεργασία είναι κοινό μας συμφέρον ανεξάρτητα από πολιτικό προσανατολισμό να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων Eurosur. Εισηγητής ο Γιάν Μιούλτερ, Άλντε. Να αρχίσουμε με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μελίντα Μπάικ. Πρώτα λοιπόν η Επιτροπή ε, εκπροσωπείται και το Συμβούλιο θα λάβουν λοιπόν ε, το λόγο Επιτροπή, Συμβούλιο και μετά εισηγητής και μέλη. Παρακαλώ κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής. Ευχαριστώ καλημέρα. Με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω σύντομα αυτή την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον ε, περασμένο Δεκέμβριο για ένα κανονισμό που να θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης συνόρων, Eurosur. Στόχος του Eurosur είναι να ενισχύσει την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων και χερσαίων σύνορων της Ένωσης. Η πρόταση αυτή είναι το αποτέλεσμα τεσσάρων ετών έντονης προπαρασκευαστικής εργασίας στην μελέτη επιπτώσεων που κάναμε. Θα δείτε μια συνόψιση των ε, όρων αναφορά στις ε, συναντήσεις ε, εμπειρογνωμόνων που προπαρασκεύασαν το κείμενο αυτό η μελέτη επιπτώσεων. Τονίζει ότι η έλλειψη μια κοινή ρυθμιστική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στον τομέα τη επιτήρηση των συνόρων, ιδιαίτερα στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, σημαίνει ότι γίνονται παράνομε ε, είσοδοι στην ε, επικράτεια τη Ένωση και εγκλήματα. Και επίση το απαράδεκτα υψηλό ποσοστό θανάτων των, πολιτών, των ε, μεταναστών που πνίγονται στα σύνορά μα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν οι αρχές της Ένωσης που ασχολούνται με τον τομέα αυτό να ε, ε, ανταλλάσσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη λειτουργία για να αποφευχθεί το έγκλημα, η παράνομη μετανάστευση και να προστατεύσουν και να σώσουν τις ζωές των μεταναστών. Η πρόταση αυτή προβλέπει το Eurosur να αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2013. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε, να εφαρμόσουμε, να ελέγξουμε και να νομοθετήσουμε ταυτόχρονα. Έτσι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να λειτουργούμε πολύ εύκολα, αλλά όλα αυτά θα είναι πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες συμπραγμαμένου του Κοινοβουλίου. Πώς λοιπόν θα λειτουργεί το Eurosur. Θα είναι μια, ένα αποκεντρωμένο σύστημα συστημάτων που θα συνδυάζει συστήματα και θα προωθεί τις ροές ε, ε, λειτουργιών θα προσπαθούμε να περάσουμε από το απλώ να κάνουμε περιπολίες στο να ανταλλάσσουμε πληροφορίε που θα σα επιτρέπουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ανταλλάσσοντα πληροφορίε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εγκληματικά δίκτυα τα οποία είναι πολύ ευέλικτα και αλλάζουν τρόπου λειτουργίας μέσα σε εβδομάδες, ενώ εμείς ε, βραδιπορούμε. Το Eurosur πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Το Eurosur θα είναι ένα σύστημα με πολλέ λειτουργίε θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, αλλά και το διαμεθοριακό έγκλημα, για παράδειγμα τη διακίνηση ναρκωτικών. Γιατί είναι οι ίδιε μέθοδοι και τα ίδια, ε, οι ίδιοι εγκληματίε οι οποίοι κάνουν αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, οι Ισπανικέ αρχέ μπορεί να αντιμετωπίζουν ε, μετανάστε οι οποίοι προσπαθούν με ένα μικρό σκάφο να περάσουν στι Ισπανικέ ακτέ και κάνουν μια επιχείρηση για να του βρουν και να του διασώσουν. Αλλά στόχος στην ουσία αυτού του αργού σκάφου είναι να απασχολήσει την ακτοφυλακή ούτω ώστε πολύ πιο ταχύπλοα σκάφη να μεταφέρουν ναρκωτικά. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε τους ε, μετανάστες που προσπαθούν ε, θαλασσίως να εισέλθουν στην Ένωση και γι' αυτό αυξάνονται κατά πολύ θάνατοι. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι 1.500 άτομα ε, πνίγηκαν πέρυσι προσπαθώντα να διασχίσουν την Μεσόγειο και η Ισπανική Guardia Civil θεωρεί ότι 6 με 10 10.000 ε, παράνομοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια και προσπαθούν να φτάσουν στα Κανάρια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη απώλεια ζωών των παρανόμων μεταναστών. Το Eurosur θα προσπαθήσει σταδιακά να βελτιώσει την συνειδητότητα της κατάστασης και την δυνατότητα αντίδραση των κρατών μελών και του Frontex και θα επιχειρήσει να εισαγάγει το νέο στοιχείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Τι σημαίνει αυτό. Τα κράτη-μέλη και το Frontex θα αποτιμούν από κοινού και συνεχώς πώς μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά. Ως παράδειγμα, αυτό θα σήμαινε ότι όταν φτάνουν σκάφη μετανάστες, για παράδειγμα στην Λαμπεντούζα, θα μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε νωρίτερα. Όλα αυτά θα επιτευχθούν βελτιώνοντα ε, ουσιαστικά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα τους δορυφόρους και τις εικόνες από τους δορυφόρους ραχοκοκαλιά θα είναι οι εθνικές αρχές συντονισμού στα κράτη-μέλη. Αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, τον Οκτώβριο του 2013 για την ανατολική και νότια περιοχή συνόρων του Σέγγεν και τον Οκτώβριο του 2014 για όλα τα ε, σύνορα Σέγγεν, χερσαία και θαλάσσια. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Eurosur θα είναι να μπορέσουν τα, κράτη, τα κέντρα εθνικής ε, προσπάθειας συντονισμού να διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών με όλες τις αρχές της χώρας που είναι αρμόδια για την επιτήρηση των συνόρων τη. Αυτό μπορεί να είναι ε, μεθοριακή φρουρή, αστυνομία, η ακτοφυλακή, το ναυτικό. Για την Eurosur λοιπόν η Ιταλία πρόσφατα ίδρυσε Εθνικό Κέντρο Συντονισμού όπου συμμετέχουν ε, οι εκπρόσωποι από τις διάφορες Ιταλικές αστυνομίες και την ακτοφυλακή και το ναυτικό. Τι ρόλο θα παίξει ε, η υπηρεσία Frontex. Στόχος της είναι να δίνει υπηρεσίες στα εθνικά κέντρα Στονισμού να παρέχει ε, προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε τα διάφορα τμήματα της Eurosur να συντονίζονται. Θα διασφαλίσει την τεχνική διοίκηση του δίκτυου της Eurosur, ούτως ώστε να υπάρχει ε, ασφαλής ανταλλαγή προφοριών το δίκτυο αυτό θα ανταλλάσσει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις περιπολίες και τα επεισόδια και περαιτέρω πληροφόρηση που θα προκύπτει από ανάλυση των εθνικών ε, καταστάσεων και την ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης. Το Eurosur δεν θα ανταλλάσσει λοιπόν πληροφορίες, αλλά θα συλλέγει και πληροφορίες. Και συνεργαζόμενοι η Eurosur και με άλλες υπηρεσίες, καθώς και με τη Frontex, θα παρέχει τα ε, όργανα για την κοινή επιτήρηση των συνόρων. Αυτή η υπηρεσία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμπεριλάβει και το ε, καθεστώς και το δίκτυο επιτήρησης των σκαφών, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε αν κάποια σκάφη, κάποια καράβια στις ε, ανοιχτές θάλασσες έχουν μια περίεργη συμπεριφορά, για παράδειγμα να προσεγγίζονται για να ανταλλάσσουν μετανάστες γνωρίζοντα ε, τι συμβαίνει στα εξωτερικά μα σύνορα, δεν επαρκεί εάν δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και ανάλογα. Προτείνουμε λοιπόν η Frontex μετά διαβούλευση με τα κράτη-μέλη να ε, καθορίζει τι επίπεδο δράση πρέπει να υπάρχει σε κάθε περιοχή συνόρων. Για παράδειγμα, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, ανάλογα με την ανάγκη αντίδραση. Οπότε τα κράτη-μέλη, συνεργαζόμενοι με τη Frontex, θα μπορούσαν μετά να κάνουν όλα τα αναγκαία για να μειωθεί το επίπεδο αντίδραση που χρειάζεται. Να βελτιωθεί δηλαδή η κατάσταση. Θεωρούμε το συνολικό κόστος για τη δημιουργία της Eurosur για την περίοδο 2011-2020 θα είναι περίπου 338 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τις νέες προοπτικές, στις νέες προοπτικές θα συμπεριληφθούν 2,44 εκατομμύρια. Κυρίως ε, θα έχουμε τον προβλημό της budget καθώς και θα έχουν, τις Frontex, συγγνώμη, καθώς και μελλοντικού πόρους που θα αποδοθούν στο μέλλον. Σας έχουμε ήδη εξηγήσει στο παρελθόν πώς θα γίνει ακριβώς η χρηματοδότηση. Τέλος, όπως είπα και νωρίτερα, για να λειτουργήσει του χρόνου, τον Οκτώβριο, το Eurosur πρέπει να κάνουν πολλά τα κράτη-μέλη, είναι μεγάλη πρόκληση και για τη Frontex. Και βεβαίως 16 από τα 18 κράτη-μέλη θα μπορέσουν να έχουν το Eurosur και έχουν ήδη δημιουργήσει τα εθνικά τους ε, κέντρα συντονισμού, η Frontex ε, εξετάζει τον τρόπο απόδοσης κονδυλίων. Κάνουμε αναλυτική αντιμετώπιση του τι θα κάνουμε το 2012 και το 2013, τους ώστε να διαπιστώσουμε σε τι βαθμό η Frontex μπορεί να καλύψει με βάση τα υπάρχοντα κονδύλια τις ανάγκες του Eurosur και σε τι βαθμό θα χρειαστούν νέες πιστώσεις και νέο ανθρώπινο δυναμικό και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση και την πρόταση. Αυτό το κοινοβούλιο το ζητούσε εδώ και καιρό κάτι τέτοιο. Από τότε που ξέσπασε ή σημειώθηκε η Αραβική Άνοιξη. Δεν είμαι βέβαια αν εκπροσωπείται εδώ και το Συμβούλιο, δεν είδαμε κανέναν. Ο κύριος Μούλτερ θα πάρει τώρα το λόγο και μετά θα δούμε αν έρθει κανείς, αν καταφτάσει κανείς από το Συμβούλιο. Ορίστε κύριε Μόλντερ μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο, και εγώ δέχομαι την πρόταση αυτή της Επιτροπής ευχαρίστως. Είναι σωστό νομίζω να υπάρχει η Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, αλλά να προσέξουμε και το θέμα των εξωτερικών σύνορων η συλλογή πληροφοριών, οτιδήποτε μας βοηθάει να μαθαίνουμε πώς θα γίνει καλύτερα των συνόρων είναι κάτι το θετικό. Η αρχή αυτή εθνικών συντονιστικών κέντρων μου φαίνεται σωστή και η μόνη μου αμφιβολία είναι ότι οι περισσότερες χώρες μέλη προβλέπουν αυτή τη στιγμή περικοπές και μέτρα λιτότητας Κατάλαβα ότι θα ζητηθεί χρηματοδότηση και από ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορέσουν να προσφέρουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Επίσης, νομίζω ότι οι ανταλλαγές εμπειριών από και πληροφοριών μεταξύ εθνικών δημοσίων υπαλλήλων είναι κάτι θετικό γιατί κάθε χώρα μέλος μπορεί να βοηθηθεί από την εμπειρία άλλης. Επομένως, συμφωνώ με την Κομισιόν ότι είναι απαράδεκτο να χάνουν τη ζωή τους τόσο πολλοί άνθρωποι στη Μεσόγειο λόγω των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, τι συνεργασία προβλέπετε μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Ξέρω ότι μερικές εθνικές αρχές και εκτός Ένωσης έχουν προσπαθήσει ή έχουν ζητήσει συντονισμό των προσπαθειών. Δεν ξέρω αν θα αρκούσε κάτι τέτοιο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί η κατάσταση αυτή τόσων απολειών ζωής. Για την προστασία των δεδομένων Βλέπω ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, δεν ζητάει πολύ προσωπικό για τη δουλειά αυτή, αλλά θα ήθελα και αυτό να επαληθευθεί κατά πόσον γίνεται δηλαδή επαρκώς αυτή η επαλήθευση. Πάντως η καλύτερη συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης είναι απαραίτητη αυτά τα κέντρα ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να πραγματοποιήσουν τέτοια συνεργασία αφού έχουμε ενιαία εξωτερικά σύνορα εδώ στην Ένωση. Προσδοκώ λοιπόν στη συνεργασία με όλους εδώ στην Επιτροπή ώστε η πρόταση τελικά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους Έφτασε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου τον οποίο καλωσορίζουμε και τον παρακαλούμε να μας φωτίσει ως προς το τι συζητάει, που έχει φτάσει το θέμα στο Συμβούλιο. Ορίστε κύριε Γιάπα Βίνκαλ Μπέτερσεν, αν το είπα σωστά το όνομά σας. Σας κατευχαριστώ για το καλωσόρισμά σας. Με συγχωρείτε που έφτασα με κάποια καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας πληροφορήσουμε για το πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο ως προς αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, συζητιέται το θέμα από το εναρμόδια ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο, προχωράει η τεχνική της εξέταση και αναμένουμε να τελειώσει η διαδικασία, η πρώτη ανάγνωση δηλαδή, μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Άρα δεν αναμένουμε έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο για αυτή την Προεδρία, αλλά από την επόμενη. Αλλά προχωράνε τα πράγματα, προχωράνε. Και Επίσης περιμένουμε την έκθεση του εισηγητή. Αυτά είχα να σας πω. Φυσικά, αν υπάρξουν απορίες, θα τις απαντήσω με τα χαράς. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα πράγματα ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις γίνουν υπό Προεδρία. Ευχαριστούμε ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος Σκούρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κείμενο που έχει προτείνει, διότι Πρόκειται για ένα κείμενο ολοκληρωμένο, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τις οποίες εμείς από καιρό έχουμε καταδείξει, θα θυμά, όπως υπενθυμίσατε κι εσείς άλλωστε, ε, βάση και λόγο των κρίσιμων καταστάσεων που ε, προέκυψαν μετά την Αραβική Άνοιξη. Είναι σημαντικά όσα υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το πεδίο της ε, ανακοίνωσης ε, να βελτιώσουμε ε, και την γνώση της καταστάσεων των συνόρων και τις δυνατότητες απόκρισης καθώς επίσης και με τρόπο ώστε να προλάβουμε και την παράνομη μετανάστευση αλλά και το οργανωμένο έγκλημα. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, δηλαδή την γνώση των συνόρων, νομίζω ότι όσα έχει πει και γράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαιτέρως σαφή και εξαντλητικά. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω ε, επί των δύο άλλων σημείων, κυρίως όσον αφορά την δυνατότητα αντίδρασης, ε, η οποία θα πρέπει μάλλον να αποσαφινιστεί καλύτερα, διότι πέρα από το γεγονός ότι γίνεται λόγος για την φυσική και προφανή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ακόμα και σε περίπτωση επανεισδοχής ε, δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ε, με ποιο τρόπο ε, θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία και όσον αφορά την πρόληψη επίσης δεν διακρίνουμε μέσα στο κείμενο ε, τα εργαλεία τα οποία μπορούν να είναι απο, ε, ε, αποτελεσματικά όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και όπως έλεγε και ο προλαλής δίνεται η δυνατότητα βεβαίως να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Πρέπει να υπάρξει τέτοια συνεργασία γιατί ε, και τα πρόσφατα ε, γεγονότα έχουν καταδείξει ε, την ανάγκη συνεργασίας με τις χώρες αυτές έτσι ώστε να προβλεφτούν τα φαινόμενα παράνομης μετανάστευσης και να δοθεί ε, κυρίως ε, η δυνατότητα ε, αποφυγής και πρόληψης της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Λέγω λοιπόν ότι χρειάζονται κάποιες διευθετήσεις, αλλά βεβαίως μπορούν να συνεργαστούν το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν επ' αυτού τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέντσιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για την εργασία που έκανε. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το οποίο μελλοντικά θα εφαρμοστεί θα συμβάλλει στο στόχο που έχει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων. Επομένως, ε, εγώ θετικός διάκειμε όσον αφορά την πρόταση αυτή. Όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά πέρα από το σύστημα Eurosur ε, και αναφερόμενες και σε όλα τα μελλοντικά συστήματα ελέγχου και επιτήρηση των συνόρων. Η διαχείριση του χώρου Σέγγεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαναδιατυπώσει πρώτα απ' όλα ε, την διακυβέρνηση του χώρου ε, Σέγγεν και μετά να εγκρίνει, να προωθήσει νέους μηχανισμούς αξιολόγησης. Χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς όλο τούτο το σύστημα Eurosur το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή και μας προτείνεται και πιθανόν ε, θα ε, εφαρμοστεί, ε, θα, δεν θα μπορέσει να είναι πλήρως αποτελεσματικό θα πρέπει να δούμε πώς προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα ε, στα πλαίσια του χώρου Σέγγεν. Δεν θα έχουμε τα μέσα και δεν θα έχουμε την δυνατότητα ε, να αντισταθμίσουμε ε, τις ελλείψεις που θα παρουσιαστούν. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτή την προβληματική της λειτουργίας των συνόρων. Εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να παρέμβουμε στις διαπραγματεύσεις με τρόπο ουσιαστικό έτσι ώστε να τροποποιηθούν κάποια τμήματα του Σέγγεν. Επανερχόμενος τώρα στη σημερινή πρόταση, θα, έλεγα στην, θα, υποβάλω μια σειρά ε, προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και άλλωστε θεωρώ ότι και η Επιτροπή μας έχει επιλέξει μια σωστή κατεύθυνση. Το θέμα των ε, ε, συνόρων. Φαντάζομαι ότι τα σύνορα θα μοιραστούν ε, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας. Τώρα, εάν τι συμβαίνει αν υπάρχει μια περιοχή, μια ζώνη η οποία θεωρείται χαμηλού κινδύνου και ξαφνικά η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, απρόβλεπτες δυσκολίες. Ε, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι δυσκολίες αυτές. Με ποια δυνατότητα παρέμβασης μπορούμε να προχωρήσουμε. Στο άρθρο 2.1 επίσης προβλέπεται ότι τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα ε, δημιουργηθούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ε, στα κράτη της Ανατολικής, της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης. Ε, ποιο είναι ποια είναι η επιχειρηματολογία, γιατί δεν θα δημιουργηθούν ταυτόχρονα όλα τα κέντρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία θα πάρει το λόγο τώρα. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που μας έδωσε ε, πληροφορίες σχετικά με το Eurosur. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό που με απασχολεί και με προβληματίζει όμως κυρίως σε σχέση με την επικουρικότητα δηλαδή είναι ασαφής η θέση της Επιτροπής δεν είναι καθόλου λοιπόν σαφής η θέση. Ε, δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια σε σχέση ε, με το τι θα γίνει αν τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν ε, να καλύψουν τις προβλεπόμενες ευθύνες τους. Επίσης, η κατανομή των πόρων και της χρηματοδότησης αναφέρεστε σε ενίσχυση και ενδυνάμωση των αρμοδιοτήτων της Frontex μέσα στα πλαίσια βεβαίως της επικουρικότητας πρέπει, να βρούμε συνολικές λύσεις βεβαίως, αλλά ο τρόπος είναι πώς θα το κάνουμε αυτό. Είναι πολλές οι χώρες οι οποίες προβληματίζονται σε σχέση με την επικουρικότητα. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Κομισιόν, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Άλμπρεχτ. Και έχουμε και άλλους έξι ομιλητές. Κύριε Άλμπρεχτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς η κυρία Κέλλες και η συγκήτριά μας, δεν είναι παρούσα, αλλά ως πράσινη έχουμε κάποιες ε, ανοιχτές ερωτήσεις για αυτή την πρόταση κανονισμού για το Eurosur. Καταλαβαίνω πολλά που ανέφερε και ο εισηγητής, διότι για πολλά θέματα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα, Χρειάζεται οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα. Το θέμα είναι αν με τα μέτρα αντιμετωπίζετε πραγματικά το πρόβλημα. Σε πολλά σημεία δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα οι κανόνοι για τη γύρω σου, τι καθήκοντα θα έχει. Για παράδειγμα, το θέμα των αποστολών εξέβρεσης και διάσωσης. Πώς θα διασώζονται τα άτομα αυτά τα οποία κινδυνεύουν ε, στη Μεσόγειο. Στην πρόταση κατά τη γνώμη μου δεν αναφέρεται. Η συνεργασία με, τρίτα, με τρίτες χώρες και μάλιστα και σε διμερές επίπεδο μεταξύ κρατών μελών και κάποιων κρατών μελών αναφέρεται με μη διαφανή τρόπο. Είναι ασαφές λοιπόν τι συγκεκριμένε αρμοδιότητες θα κατανέμονται μεταξύ αυτών των ε, συνεργαζομένων και με ποια νομική βάση θα γίνονται όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια βασική ασάφεια. Ποια σχέση θα υπάρχει μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των διαφόρων αρχών εφαρμογής του δικαίου. Ποιος θα κάνει τι δηλαδή εφόσον ε, τίθεται θέμα διαφάνειας, θεωρώ ότι λείπει σε πολλά σημεία η διαφάνεια. Καθώς και δεν είναι σαφές ποιος θα έχει την πολιτική ευθύνη και τον πολιτικό έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά δεν ε, περιγράφονται επαρκώς, κατά τη γνώμη μου, στο κείμενο, το θέμα της προστασίας δεδομένων. Δεν ε, είναι σαφές για μένα η επεξεργασία των ε, ηλεκτρονικών στοιχείων από τη Γύρω σου δεν περιχαρακώνεται σαφώς. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω ε, δυνατότητες ανταλλαγής στοιχείων. Ήδη υπάρχουν ε, υπηρεσίες που το κάνουν. Η Europol θα έπρεπε να είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος όπως είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως μπορεί να συμπεριληφθεί και η Frontex, αλλά σε αυτό το κείμενο δεν καθορίζονται αυτά τα πράγματα. Και τελευταίο, ήδη αναφέρθηκε, μελέτη των επιπτώσεων και θέμα επικουρικότητας. Χρειάζεται να διευκρινιστούν αυτά αν πρόκειται να δαπανίσουμε τόσα χρήματα για αυτό το θέμα. Ενώ δεν είναι σαφές τι τελικό αποτέλεσμα θα έχουν, πώς θα αξιοποιηθούν, πώς θα συμβάλλουν τα κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες. Απλώς αναφέρεται ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στις ΗΠΑ με το λεγόμενο ZipNet, που και αυτό έχει τεράστιο κόστος και το οποίο διεκόπη λόγω προβλημάτων με την μελέτη επιπτώσεων. Δεν θα είναι σκόπιμο να κάνουμε τα ίδια λάθη. Χρειαζόμαστε λοιπόν επαρκή εξέταση του πώς θα αξιοποιηθούν οι πιστώσεις και πώς θα εξαγάγουμε συμπεράσματα. Περιμένουμε λοιπόν τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δίας μέρα. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία. Δεν είναι καινούρια. Υπάρχουν προηγούμενα. Θα αναφερθώ σε αυτά. Και θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια για τις ε, ευαισθησίες που προβλέπω, για τα προβλήματα που προβλέπω. Πρώτον, ήδη στα περίφημα ΣΥΒΕ τα συστήματα ηλεκτρονικής, τα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι η αρχή της επιτήρησης ε, των νότιων συνόρων που άρχισαν να λειτουργούν από το 2002 όταν υπήρξε το πρόβλημα εισρωής παρανόμων μεταναστών. Αυτά τα σύστημα ηλεκτρονικής ε, επιτήρησης επέδειξαν ε, τις αδυναμίες τους όταν υπάρχουν, για παράδειγμα, δυσχερείς μετεωρολογικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν στα αεροσκάφη ορίων να πετάνε. Το σύστημα που μας προτείνεται, από ό,τι φαίνεται, για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, έτσι μας λέγεται, είναι ε, ανέφικτο. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν ε, όλα μας τα νότια σύνορα. Το αποδεικνύει η εμπειρία μας. Η μόνη μου ελπίδα είναι το σύστημα αυτό να βοηθήσει να σωθούν ζωές για διασώσεις. Γιατί τα στοιχεία από την Guardia Civil που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεπαρκή. Μιλήσατε για 6.000 νεκρούς στον Ατλαντικό. Συγγνώμη. Είναι, ε, είπατε 6 και 10. Περισσότερο πιο κοντά στις 10.000 από τότε που ξεκίνησε αυτή η κρίση μετανάστευσης ε, παράνομης. Με ενισχύει λοιπόν το θέμα αποτελεσματικότητας και κατά πόσον είναι ανάλογα τα μέτρα αυτά, κατάλληλα και με ανισχύει και το θέμα του κόστους. Το πιο θετικό που μπορεί να προκύψει πέρα από τον έλεγχο των συνόρων, δηλαδή ανεξάρτητα από τον έλεγχο των συνόρων, είναι να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν περάσει κάποια θαλάσσια σύνορα για να μπορέσουμε να τους σώσουμε. Όσον αφορά τα στοιχεία του συστήματος, συντονισμός της ανταλλαγής ροών πληροφοριών και επεξεργασμένων πληροφοριών. Το πιο αποτελεσματικό που θα μπορούσε να διαρκέσει είναι η επεξεργασία των πληροφοριών για να μας επιτρέψει να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Και η πληροφόρηση απλή θα βοηθήσει μόνο τη διάσωση. Τα κέντρα συντονισμού, κατά τη γνώμη μου, έχουν ήδη λειτουργήσει. Υπάρχουν προηγούμενα. Από το 2002, όταν ε, προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα που το λέμε Fuerteventura. Στο Fuerteventura και άλλο στα στενά. Και το τρίτο που δεν νομίζω ότι άρχισε να λειτουργεί γιατί υπήρξαν διαφωνίες για το πώς θα λειτουργήσει. Νομίζω πως είναι καλό το σύστημα αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον τίτλο του που είναι επιτήρηση των ε, συνόρων. Πώς να επιτηρήσεις τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Αναμένουμε λοιπόν όλοι τα σχόλια όλων μας ε, για να τα λάβει υπόψη ε, ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα θεμελιώδη θέματα που θέσατε. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ δέχομαι την πρόταση αυτή γιατί νομίζω θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ακριβέστερη γνώση της κατάστασης στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά και γιατί νομίζω ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη βελτίωση της εργασίας του Frontex, μετά μάλιστα από την αναθεώρηση της εντολής του. Έχω όμως και μερικά σχόλια που θέλω, για ερωτήματα που θέλω να θέσω στην Κομισιόν και ελπίζω να είναι σε θέση να μου απαντήσει. Πρώτον, προβλέπει ή όχι καμία καινούρια υποδομή για την εφαρμογή του Ευρωσούρ ή αντίθετα προβλέπει το συνδυασμό των υπαρχουσών υποδομών από τα διάφορα κράτη-μέλη και το συντονισμό θα χρησιμοποιηθεί τελείως καινούργια τεχνολογία ή απλώς θα συνδυαστούν τα υπάρχοντα. Δεύτερον, όλοι γνωρίζουμε ότι από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την εποπτεία ή επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων είναι η ταύτιση των μικρών πλοίων πλοιαρίων είναι σαν να ψάχνουμε βελόνα στον αχυρόνα η καρφίτσα. Αυτό το καινούργιο, αυτή η καινούργια πρόταση λοιπόν θα μπορέσει ή όχι να λύσει το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ένταση όλη την τελευταία δεκαετία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε έτσι ευκολότερα να ταυτίζουμε τα προβληματικά πλοιάρια που είναι η μεγαλύτερη πηγή απώλεια ζώων ενώ παράλληλα οι, αυτοί που οργανώνουν τη λαθρομετανάστευση έχουν τεράστια έσοδα. Τρίτον, για τις ανταλλαγές πληροφοριών και δεδομένων, από ό,τι γνωρίζω εγώ, το Ευρωσούρ αφορά την περιγραφή ολόκληρων καταστάσεων και όχι προσωπικά δεδομένα. Άρα δεν θέτει το Ευρωσούρ κανένα θέμα συλλογής ή ελέγχου προσωπικών δεδομένων. Μπορεί όμως να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο εφόσον τεθεί το θέμα της ανταλλαγής προσωπικών. Για τις τρίτες χώρες τώρα Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη ε, έχουμε την, τις ροές από τη Βόρεια Αφρική και ότι εκεί στις χώρες της Βόρειας Αφρικής υπάρχει μεγάλη έλλειψη υποδομών και επιτήρησης. Ξέρουμε ότι μεγάλοι αριθμοί πλοιάριων φεύγουν αυτή τη στιγμή από τη Λιβύη ενώ προηγουμένως η ροή ήταν προς την αντίθετη πλευρά, προς τον νότο και την έρημο. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν τις τρίτες χώρες να δημιουργήσουν δικές τους υποδομές που να τις συνδυάσουν, να τις συνδέσουν με την Ευρωσούρ. Χρειάζεται συνεργασία και μεταξύ των τρίτων χωρών και συνδυασμός της με του Ευρωσούρ. έπειτα το κόστος. Αν κατάλαβα καλά η Κομισιόν προτείνει 338 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Μπορείτε να μας πείτε πού θα διατεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Αν πρόκειται να διατεθούν σε ανθρώπινους πόρους, σε νέα τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε εδώ περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κόστος που προβλέπετε. Απ' την άλλη είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί η Ιδανική Προεδρία ήδη παρετείται και λέει ότι θα λυθεί το θέμα από την Κυπριακή. Επειδή είναι τόσο σημαντική η πρόταση, νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτερα. Αν πράγματι θέλουμε από την 1η Οκτωβρίου να ισχύσει αυτό το ευρωσούρο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον εισηγητή κύριο Μούλτερ που ελπίζω να μας οδηγήσει σε θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω και εγώ στο τέλος την Προεδρία πώς θα μπορούσε να επιταχύνει ο κύριος Μπρόντς και μετά και άλλοι, αλλά και άλλες. Ακούσαμε τους τρομακτικούς αριθμούς των χιλιάδων μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους, λάθρων μεταναστών. Και ακούσαμε επίσης ότι θα γίνεται καλύτερη επιτήρηση. Πώς θα αντιδράσουν σε αυτό, αν τους επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση και τους χορηγηθεί ακόμη και καθεστώς ε, ασύλου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο για να λαθρομεταναστεύσουν. Αν η απώλεια των ζώων θέλουμε να αποτραπεί, τότε οι είσοδοι στην Ένωση πρέπει να ελέγχονται καλύτερα, με ή χωρίς συνεργασία των υπολείπων χωρών. Όσοι φτάνουν στην Ευρώπη δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα διαμονής αυτομάτως. Αν μας ενδιαφέρει η απώλεια της ζωής πρέπει να μιλήσουμε και για τα ναρκωτικά. Γιατί οι περισσότεροι λατρομετανάστες προέρχονται από τις χώρες από που προέρχονται και τα ναρκωτικά. Το πρόβλημα λοιπόν δεν περιορίζεται στα λιμάνια της Βόρειας Αφρικής αλλά γενικότερα στα νότια σύνορα και των χωρών αυτών της Βόρειας Αφρικής από όπου τα ναρκωτικά. Ξέρω ότι οι φίλοι του κυρίου Σαρκοζή και του κυρίου Κάμερον υποτίθεται ότι με τους βομβαρδισμούς τους έφεραν τη δημοκρατία και την ειρήνη στη Λιβύη, αν και μάλλον αφορούσε το πετρέλαιο παρά την ειρήνη και τη δημοκρατία η επιχείρησή τους. Κυρία Σίπα. Ευχαριστώ ήδη. Υπόθηκαν ορισμένα για τους βασικούς στόχους, αλλά και για τα ενδεχόμενα προβλήματα αυτού του σχεδίου να θέσω ένα θεμελιώδες θέμα και μόνο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουμε την, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Όμως έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το επιτύχουμε. Είτε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και εφαρμογή θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη τα ίδια στα εξωτερικά σύνορα. Ερώτημα. Μήπω η προστασία των εξωτερικών σύνορων δεν θα έπρεπε να είναι κοινοτικό καθήκον. Ακόμη και τα κράτη-μέλη δηλαδή που δεν έχουν εξωτερικά σύνορα να συμμετέχουν. Ερώτηση λοιπόν. Υπάρχουν σκέψει προ αυτή την κατεύθυνση. Να συμμετάσχουν και κράτη όπω η Γερμανία οικονομικά, τεχνικά ή με προσωπικό στην προστασία των εξωτερικών σύνορων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε. γιατί αλλιώ θα πρέπει να έχουμε συνεχώ αυτέ τι ε, αναφιόμενε συζητήσει για ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Έρνστ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα σας εκπλήξει ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η πρόταση. Κατά πρώτον, βασίζεται σε ένα μεγάλο σφάλμα ότι μπορούμε ερμητικά να κλείσουμε τα σύνορά μας τα εξωτερικά. Το είπαν ήδη και άλλοι συνάδελφοι. Τέτοιοι έλεγχοι που επιδιώκονται δεν είναι δυνατόν επιτύχουν αυτό που στοχεύουν. Δύσκολα καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε αυτή την πρόταση ως ε, προστασία των ε, προσφύγων. Αυτά είναι κοινικά πράγματα. Αυτή είναι η βασική μας θέση. Δεν σας εκπλήσει νομίζω η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τρίτες χώρες ε, θεωρώ ότι είναι εντελώς ε, ασαφής. Δεν ρυθμίζεται παρκώς, μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Γιατί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να τεθεί περισσότερο ως προτεραιότητα. Βεβαίως, αυτό είναι θέμα που πρέπει να τεθεί και για την Frontex. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να επεκταθεί περισσότερο η αρμοδιότητα των συνόρων αυτών. Έθεσαν πολλοί συνάδελφοι και το θέμα του κόστου. Πρέπει να μιλήσουμε για αναλογικότητα. Αναλογικότητα των μέτρων σε σχέση με στόχους που κατά τη γνώμη μου ποτέ δεν θα επιτευχθούν. Θέτω λοιπόν το ερώτημα ποιος θα πληρώσει αυτά τα μέτρα. Είναι λάθος να περνάμε από τη μία πρόταση στην άλλη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων πριν να εξετάσουμε πώς έχει όντως η κατάσταση, πώς θα την αντιμετωπίσουμε και πώς θα τη συνδυάσουμε με την προστασία των προσφύγων που για καλούς λόγους, για σωστούς λόγους θέλουν να μπουν στην Ευρώπη. Φρούριο Ευρώπη, να το πω σαφές, σαφώς, δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτή λοιπόν η πρόταση της Επιτροπής θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα λαθασμένα. εκφράζω μεγάλες επιφυλάξεις έναντι αυτής της προτάσεως. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιακολίνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή θα δώσει πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ε, του 2013. Έχουν προβλεφθεί επιπλέον πόροι όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Επομένως, ερώτηση, εάν όντως αυξηθούν 40% οι πόροι και εάν επίσης είναι γεγονός ότι το κόστος το οποίο συνδέεται με την ενεργοποίηση και λειτουργία του ε, Eurosur προβλέπουν 338 εκατομμύρια ευρώ, αυτά ε, τα επιπλέον κονδύλια προφανώς θα αφορούν την δραστηριότητα Eurosur. Είναι λοιπόν μια προστιθέμενη αξία. Ε, ε, θα πρέπει δηλαδή η Eurosur να έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Δεν ξέρω επίσης εάν θα δημιουργηθούν νέες υποδομές ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες. Ποια προσέγγιση, ποια σχέση δυνάμεων θα έχει αυτός ο οργανισμός με άλλους οργανισμούς ξεκινώντας από την Frontex. Τι είδους συντονισμός μπορεί να προβλεφθεί επίσης σε σχέση με δραστηριότητες τρίτων χωρών, γιατί εδώ λαμβάνεται υπόψη και η μεσογειακή, ε, η μεσημβρινή διάσταση της ε, Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου στην ε, Μίνη Ολομέλεια θα μιλήσουμε για τη Λαμπεντούζα. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο η Eurosur μπορεί να κάνει την Ευρώπη πιο αποτελεσματική, πιο, ε, ε, πιο γενναιόδορη αλλά και πιο αλληλέγγυη απέναντι στην κατάσταση έτσι όπως αυτή διαγράφεται. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος πραγματικά να δώσει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Πάικα έτσι ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα στο μέτρο του δυνατού βεβαίως, γιατί ετέθησαν πάρα πολλά προβλήματα, ανησυχίες και ερωτήματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έθεσαν ερωτήματα. Ε, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ, να αποκριθώ μάλλον στα κύρια ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Έτσι ώστε να μάθουν και κάποια πράγματα επιπλέον τα μέλη της κοινοβουλίας. Το Eurosur δεν είναι, είναι ένα εργαλείο, ένας μηχανισμός ε, ε, στρατηγικής και δεν ε, αφορά άλλες διαδικασίες όπως είναι ο χώρος έγκαινε, ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών κτλ. Βεβαίως θα υπάρξει συνεργασία και βεβαίως υπάρχουν συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το ευρύτερο ζήτημα της βελτίωσης του Σέγγεν εξακολουθεί να λαμβάνει η χώρα. Εδώ αναφερόμαστε σε διαχείριση συνόρων. Ε, να πω δύο λόγια όσον αφορά το κόστος. Έγινε αναφορά στην εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως εμείς ε, προσπαθήσαμε να δούμε τα συστήματα, τα παρόμοια συστήματα τα οποία λειτουργούν απανταχού ε, του κόσμου. Το 10% το δικό μας κόστος αφορά περίπου το 10% των 3,5 περίπου ε, εκατομμυρίων που έχει δώσει, έχει δαπανίσει και προβλέψει να δαπανίσει ε, να δαπανίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, επίσης, εμείς προσπαθούμε να βρούμε τις βέλτιστες ή τις μη βέλτιστες πρακτικές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε σχέση με το κατά πόσον τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεσμεύσουν τα απαραίτητα ποσά, είναι ένα ζήτημα βεβαίως το οποίο ε, θα προκύψει στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη πάντως ήδη ε, δίνουν πολλά χρήματα για την διαχείριση των εξωτερικών τους ε, συνόρων και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική η καλή συνεργασία. Στην, ε, ε, επίσης ε, έχουμε και την επόμενη εβδομάδα συνάντηση της ομάδας εργασίας για τη δεύτερη ανάγνωση για τα σύνορα ISF και το θέμα θα συζητηθεί και στην ομάδα αυτή. Οι σχέσεις τώρα με τρίτες χώρες και συμφωνίες με τρίτες χώρες. Προφανώς στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση στις γειτονικέ χώρες, ε, χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κύματα των ε, μεταναστών και βεβαίως αυτή Αυτά έχουν ήδη προβλεφθεί ε, στην πρόταση για τη συνολική μετανάστευση και, την, ε, και τις μετακινήσεις των ε, πληθυσμών. Επίσης, θέλουμε να καταδείξουμε ότι υπάρχουν προβλέψεις για ειδικά τμήματα των συνόρων τα οποία αντιμετωπίζουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ιδιαίτερο βάρος ή ιδιαίτερα προβλήματα αυτό βρίσκεται στο άρθρο 15.1c, όπου αναφέρεται σαφώς ότι και το Εθνικό ε, Κέντρο Συντονισμού θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον στήριξη από την ε, Frontex. Στήριξη η οποία θα προέρχεται μετά από και θα αποφασίζεται μετά από συντονισμένη προσέγγιση των προβλημάτων. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή ε, του, ε, αν θα γίνει δηλαδή τον Οκτώβριο του 2013 και τον Οκτώβριο του 2014. Αναγνωρίζουμε ότι έχει γίνει ήδη πολλή ε, δουλειά ε, έτσι ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί η EuroSource. ε, βεβαίως πολλή προσπάθεια απαιτείται και από πλευράς της Frontex και από πλευράς των κρατών μελών. Τώρα, τα ζητήματα τα οποία θίγησαν ε, σχετικά με τις ε, ε, επιχειρήσεις διάσωσης τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να δώσουν προτεραιότητα ε, στην διάσωση, στην αναζήτηση και την διάσωση. Ε, και αυτό βεβαίως και σύμφωνα με, την, ε, με, τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες της του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και το, κυρίως το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην διάσωση στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, η Eurosur δεν αμφισβητεί ε, την, ε, ε, τις δικαιοδοσίες των ομάδων διάσωσης και άλλωστε και η απόφαση 2010 για τις κοινέ προσπάθειες και επιχειρήσεις διάσωσης δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και αυτό αναφέρεται ρητά και στην αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 13. Επίσης αναφέρεται ρητά ότι η Eurosur δίνει προτεραιότητα στη την διάσωση των ζώων των ε, μεταναστών. Άρθρο 19, σημείο ε. Όσον αφορά τώρα την προστασία των δεδομένων ε, και στην, ε, στο επεξηγηματικό μνημόνιο αναφέρεται ότι δεν θα χρησιμοποιούνται ε, στοιχεία προσωπικού ε, χαρακτήρα, αλλά ε, θα ανταλλάσσονται πληροφορίες για απρόσωπα στοιχεία, όπως ας πούμε αριθμός δίωξη σκαφών, περιστατικών που εμπλέκουν, συμβάντων που εμπλέκουν σκάφη κτλ. Βεβαίως, ο τροποποιημένος κανονισμός Frontex δίνει τη δυνατότητα στην Frontex σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις αξιολόγησης κινδύνου κυρίως ε, δίνει τη δυνατότητα, λέω, στη Frontex να ανταλλάσσει ε, κάποια στοιχεία προσωπικού δεδομένου στο προήμιο, όμως εδώ αναφέρεται ότι οπωσδήποτε αυτού του είδου η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ε, θα συμμορφούνται απολύτως με τα όσα προβλέπονται από τις, από τις Εθνικές Νομοθεσίες Προστασίας των Δεδομένων και θα διέπονται και από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά τώρα την επικουρικότητα. Με μεγάλη προσοχή έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό βεβαίως. Ε, ε, στα χέρια των κρατών μελών βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθύνη όπως και τώρα. Ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Frontex ε, λειτουργεί ε, σαν ε, παροχές υπηρεσιών και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να διαραγεί ή δεν υπάρχει πρόθεση διάρρηξης της αρχής της επικουρικότητας. Επίσης, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανείχνευση των ε, των ε, σκαφών τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επίσης ε, είναι δύσκολος ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων στις μελλοντικές διομοσιονομικές προοπτικές γίνεται σαφής αναφορά στα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να σας πω ότι έχει υπάρξει χρηματοδότηση και, από, και, ε, και ε, όσον αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού ε, το, στις τρίτες χώρες. Τώρα, το πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα, πώς ακριβώς θα δαπανηθούν, δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή αναλυτικά, αλλά πάντως τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης. Αργότερα θα υπάρξει αναλυτικότερη πληροφόρηση. Ε, και θα δώσουμε και βεβαίως τις πληροφορίες αυτές και στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα ε, να ζητήσω τον, εκπρόσωπο του Συμβουλίου, εάν θέλει να πάρει το λόγο, εάν θέλει ε, να πει δύο λόγια. Σύντομο όμω είναι δυνατόν, γιατί από ό,τι έμαθα μόλι τώρα, ο κύριο Κύρκο, ο επόμενο ηγητή, θα πρέπει να φύγει ε, το στι 12 και επομένω θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Ε, αν θέλετε να πείτε κάτι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία σύντομα να απαντήσω στον δόκτορα Μπουσούτιλ. Χαίρομαι που συμφωνεί ότι είναι σημαντική η πρόταση και ότι χρειάζεται να γίνει πρόοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος όσο το δυνατόν συντομότερα. Η Προεδρία οργάνωσε σε όλες τις, τις συναντήσεις και συζήτηση του θέματος αυτού, αλλά επειδή είναι τεχνικό το θέμα, χρειάζεται χρόνος για την εντελεχή του εξέταση. Και όπως σας είπα και πριν, η Δανική Προεδρία προσπάθησε να το τελειώσει αλλά διαβεβαιώ και τον κύριο Μπουσουτήλ και τους υπόλοιπους ότι και εμείς συμφωνούμε ότι χρειάζεται ταχεία πρόοδος αν καταστεί δυνατόν να λήξει το θέμα πριν λήξει η Προεδρία θα είμαστε και εμείς πιο ευχαριστημένοι ο εισηγητής κύριος Μούλτερ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αποδοχή της έκθεσης από τους συναδέλφους. Γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικό τα εξωτερικά μας σύνορα να τακτοποιηθούν. Ελπίζω να συνεργαστώ θετικά με όλους σας τους επόμενους μήνες για να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να είναι αποδεκτή όχι μεν για από όλους αλλά από τους περισσότερους εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείωσα όλα όσα υπόθηκαν και θα τα συμπεριλάβω στις τροπολογίες μου. Ευχαριστούμε. Δύσκολη δουλειά. Επόμενο θέμα είναι τα στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία των επιβατών. Ο κ. Κύρκο πρέπει να φύγει τώρα το μεσημέρι. αλλά και αφού φύγει θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Ελπίζω να είναι κάποιος εδώ που να δεχτεί να σας πληροφορήσει μετά για το τι θα έχει υποθεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, πάνω από 400. Παρακαλούμε λοιπόν κύριε κύρκο, συνοψίστε μας λίγο τι φρονείτε για τις τροπολογίες αυτές, όχι μία-μία βέβαια. Ορίστε. Ευχαριστώ πρόεδρε, συγγνώμη που έχω άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά το προσωπικό μου εδώ θα, θα με πληροφορήσει για ό,τι θα έχετε πει στη συνέχεια αφού φύγω. Όπως είπατε και εσείς είναι πάνω από 400 οι τροπολογίες, 300 και 489 μάλιστα τελικά. Όλες είναι σημαντικές για όσους τις συνέταξαν βέβαια. Αλλά το γεγονός ότι είναι τόσο πολλές δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον ότι πρόκειται για πολύπλοκο θέμα και το λένε και παραδέχονται πολλές από τις τροπολογίες αλλά επίσης δείχνει γιατί θα μιλήσω για τρεις-τέσσερις από τους κυριότερους που μιλούν για τους κυριότερους τομείς της έκθεσης μου δείχνει ότι πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ ως συγητής για να καταλήξω σε συμβιβασμούς και συνδυασμούς των τροπολογιών. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω βέβαια γιατί έχω και εγώ τις απόψεις μου, όπως και οι συντάκτες των τροπολογιών. Αλλά θα κάνω παρόλα αυτά ό,τι μπορώ για να πετύχω συμβιβασμούς που να απλοποιήσουν τα πράγματα και να είναι πιο εύκολη η διεκπαιρέωση της έκθεσης. Η ιδέα της δημιουργίας ενός δικού μας ευρωπαϊκού συστήματος PNR είναι ελκυστική. Ε, εδώ και μερικούς μήνες αρχίσαμε να συζητάμε το θέμα και κατέστη σαφές ότι παρά τις τροπολογίες υπάρχουν προβλήματα εκκρεμή. Πρώτον, πολλές τροπολογίες ζητούν το ευρωπαϊκό αυτό PNR να αφορά αποκλειστικά την τρομοκουρατία αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες PNR για προσωπικά στοιχεία επιβατών που προσπαθούν να απομονώσουν το ενδιαφέρον του μόνο σε αυτόν τον τομέα. Εγώ πιστεύω ότι και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα γενικότερα είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όχι μόνο η τρομοκρατία. Ορισμένοι γνώρισαν, είχαν εμπειρία τρομοκρατίας, άλλοι όχι στις χώρες μας. Και το να περιορίσουμε εδώ το θέμα στην τρομοκρατία νομίζω ότι θα ήταν απαράδεκτο για τις χώρες που δεν έζησαν με τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά έχουν εμπειρία από τα τρομερά διεθνή οργανωμένα εγκλήματα που σημειώνονται και δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως νομοθέτες για να διασφαλίσουμε ότι αν εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα δεν θα αφορά μόνο ένα θέμα όπως την τρομοκρατία. Μερικές χώρες μέλη, πρόεδρε, μέχρι και 95% των κατασχέσεων ναρκωτικών τους όπως το Βέλγιο τις οφείλουν στη χρησιμοποίηση τέτοιου συστήματος PNR και έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες μέλη και για τις συλλήψεις λαθρεμπόρων ναρκωτικών και δουλεμπόρων πέθων. Και υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να μην θεωρούνται επισήμως τρομοκρατικές, αλλά που έμεσα λόγω των χρηματικών τους επιπτώσεων καταλήγουν στη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Η Επιτροπή έχει επιτρέψει τη χρήση των υπαρχόντων συστημάτων PNR τουλάχιστον για την τρομοκρατία και οι τροπολογίες που ζητούν τον περιορισμό σε αυτό το θέμα τις κατανοώ αλλά δεν δέχομαι τον περιορισμό. Δεύτερον, το θέμα της συλλογής των στοιχείων ή των στοχευμένων πτήσεων. Είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα μεταξύ μας. Η συλλογή στοιχείων για λιγότερες πτήσεις ή με πιο στοχευμένες, πιο επικίνδυνες πτήσεις θα σήμαινε ότι μειώνουμε τον αριθμό των στοιχείων που συλλέγονται από τους επιβάτες και επιβάτησες και πιστεύω ότι ένα σύστημα που θα συλλέγει στοιχεία μόνο για τις πιο επικίνδυνες πτήσεις είναι το ίδιο επικίνδυνο διότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές των κριτήριων που θα θεωρήσουμε ως επικίνδυνες πτήσεις. Γιατί έτσι θα δημιουργούσαμε ένα σύστημα με ελλείψεις εφόσον μάλιστα η αξία του συστήματος αυτού βασίζεται σε στοιχεία που θα αξιολογηθούν εκ των υστέρων, όχι αμέσως μετά τις πτήσεις. Και έπειτα οι ορισμοί μπορεί να εξαρτώνται και από τις χώρες μέλη που θα καθορίζουν τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνη πτήση ή προορισμός. Πόσο σύντομα θα αλλάζουν τα δρομολόγια κάποιας επικίνδυνης πτήσης, αυτό δεν είναι βάσιμο. Φυσικά οι τρομοκράτες δεν ε, χρησιμοποιούν πάντα τον ευκολότερο ή τον πιο προφανή δρόμο από το α στο β με σε ευθεία γραμμή. Πάνε από το α στο ζ στο ε, ζ ε, και μετά καταλήγουν στο β. Είναι γνωστή γνωστά τα πολύπλοκα δρομολόγια που χρησιμοποιούν και οι τρομοκράτες και οι μυστικές υπηρεσίες. Κάτι άλλο αμφιλεγόμενο όπου υπάρχουν αντιρρήσεις um, και που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως εισηγητή είναι το ότι μαζί με την 100% συλλογή στοιχείων για όλες τις πτήσεις και οι εσωτερικές πτήσεις μέσα στην Ένωση πρέπει να γίνουν αντικείμενο αυτής της συλλογή πολλες πολλές. Πολλά κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Εγώ όμως νομίζω ότι είναι σωστό γιατί οι τρομοκράτες και οι οργανωμένοι εγκληματίες δεν χρησιμοποιούν πάντα δρομολόγια άμεσα ούτε τα σημειώνονται τα εγκλήματα μόνο κατά την είσοδο έξοδο στην Ένωση και μεταξύ των χωρών της Ένωσης υπάρχει, σημειώνεται οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Δεν θα ήθελα να, να φυγήσουμε ένα πλοίο που θα έχει τρύπε. Νομίζω το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες από την αρχή. Αναγνωρίζω βέβαια γιατί υπάρχουν οι αντιρρήσεις αυτές. Τέλος, τα τέσσερα σημεία που θέλω να τονίσω. Η αναγκαιότητα πρώτον. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα. Συμφωνούν οι περισσότεροι από αυτό. Όσοι πιστεύουν ότι μάλλον το αντίθετο, ότι δεν χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα, φυσικά δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Εδώ είναι θέμα και προστασίας των δικαιωμάτων και της ίδιας της ζωής των επιβατών και της ασφαλέστερης λειτουργίας των αερογραμμών και η συζήτηση αυτή γίνεται σε πολλά βήματα, αλλά και σε αυτό δηλαδή το θέμα της συλλογής πληροφοριών επιβατών μέσα στην Ένωση. Χρειάζονται σαφή κριτήρια, αλλιώς θα γίνεται μόνο διμερός η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών για τους επιβάτες, χωρίς καμία νομική σαφήνεια και βεβαιότητα. Μερικοί θεωρούν ότι η δημιουργία μίας ενιαίας τράπεζας δεδομένων είναι κάτι το θετικό, άλλοι όχι. Πρέπει η νομοθεσία να είναι σαφής ως προς την προστασία όχι μόνο των επιβατών αλλά και των κυβερνήσεων. Αυτά τα λέω διότι εδώ υπάρχουν οι διαφωνίες. Όπου υπάρχουν δηλαδή τροπολογίες που διαφωνούν μαζί μου. αλλά υπάρχουν και πολλές με τις οποίες συμφωνώ. Πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα και εγώ με τους σκιώδεις συναντιέμαι συχνά και θα συνεχίσω να συναντιέμαι. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι αποδεκτό στο τέλος ιδιαίτερα ως προς το θέμα της αποθήκευσης και διατήρησης των δεδομένων Είμαι σχετικά αισιόδοξο. Ξέρω ότι και σήμερα αργότερα θα συζητήσετε για το θέμα της απειλής που υφίσταται η Ευρώπη από το οργανωμένο έγκλημα και θα μιλήσει η Ευρωπόλ. Σημαντική και αυτή η συζήτηση. Αλλά το σύστημα που συζητάμε θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και την Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος Είμαι ευγνώμων προς την Κομισιόν, τους Σκιώδης και τους συναδέλφους και ελπίζω τώρα ότι η Προεδρία του Συμβουλίου, ότι με τις συμβιβαστικές τροπολογίες μάλλον, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ταχύτερα. Μια ομάδα ευρωβουλευτών μεταξύ τους και εγώ θα πάμε να επισκεφθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο το αρχηγείο, το συντονιστικό αρχηγείο του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για να δούμε πόσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο το σύστημα αυτό και για εκείνους. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα επίσκεψη για όσους έρθουν. Στις 31 Μαΐου προβλέπεται η ψηφοφορία, αν κατάλαβα καλά. Και μέχρι τότε θα κάνω σκληρή προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμβιβαστικό κείμενο αλλά που να αποτελεί πραγματική πρόοδο ως προς αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση που μας δώσατε όσον αφορά τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία. Πρώτα απ' όλα θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, εάν υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, να μας ε, πει τις ε, απόψεις του για τις τροπολογίες κυρίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, ο αριθμός των τροπολογιών είναι πολύ μεγάλος και θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στα κυριότερα σημεία. Υπήρξαν ε, τροπολογίες σχετικά με την μείωση του πεδίου προς δύο κατευθύνσεις. Μία ε, για περιορισμό της ε, οδηγίας μόνο σε τρομοκρατία και να αφαιθεί εντελώς, να διαγραφεί εντελώς το θέμα των εγκληματικών ενεργειών. Εμείς συμφωνούμε με τον κύριο Κέρκοπ ότι ότι αυτός δεν θα ήταν χρήσιμος τρόπος εργασίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία να χρησιμοποιείται κυρίως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, είτε πρόκειται για ε, εμπόριο ανθρώπων, είτε για εμπόριο ναρκωτικών, αλλά γενικότερα για σοβαρές εγκληματικέ πράξεις. Και επομένως θα χάναμε την προστιθέμενη αξία του συστήματος PNR εάν βγάζαμε ε, όλα τα στοιχεία που αφορούν το έγκλημα έξω από το πεδίο της οδηγίας αυτής. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες για μείωση του πεδίου και θέλουν λοιπόν αυτή η κατεύθυνση αφορά ε, την, τον περιορισμό σε ε, τρομοκρατία και ε, διαμεθοριακό έγκλημα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία του συστήματος PNR. Αυτό κάναμε εμείς τελικά και το κάναμε για τον λόγο που σας εξηγώ. Για ανείχνευση ε, ε, προσώπων, ε, εγκληματιών δηλαδή, που δεν σχετίζονται με διαμεθοριακό έγκλημα, αλλά δεν έχει έννοια να περιορίσουμε την, το πεδίο εφαρμογής μόνο στα διαμεθοριακά εγκλήματα και να αφήσουμε απ' έξω τέτοιους εγκληματίες Θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ με αυτό που συχνά αναφέρεται ως profiling. Το άρθρο 4 της πρότασης υπήρξαν πολλές ε, προτάσεις τροπολογιών για το 4. Στόχος των τροπολογιών είναι να αποκλείσουν ε, την χρήση στοιχείων PNR για την ε, πρόβλεψη κινδύνου ε, είναι κατανοητό βεβαίως ότι η έννοια της ε, διενέργειας σχεδίων ε, πρόληψης κινδύνου βάσει των στοιχείων των επιβατών είναι ευαίσθητο αλλά δεν είναι παράνομο. Η Ευρώπη αναγνωρίζει την χρήση αυτών των στοιχείων και ήδη στις συστάσεις του 2010 τις θεωρεί νόμιμες και Επομένως ε, θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επίσης όλες ε, οι προφυλάξεις ε, στην παρούσα πρόταση έτσι ώστε ε, να αποφευχθούν εγκληματικές ή παράνομες πράξεις. Επομένως δεν έχουμε πρόβλημα με την πρόταση που έχουμε υποβάλει, δεν είναι παράνομη με κανένα τρόπο, αφορά την εφαρμογή του δικαίου, βεβαίως μπορεί να είναι ευαίσθητα αλλά όχι παράνομη δεν μπορούν να αποκλειστούν αυτές τις δραστηριότητες από την πρόταση γιατί ε, πραγματικά εκεί έγκυται η σημασία και η χρήση του PNR. Ε, θα ασχοληθώ τώρα με ένα άλλο θέμα, είναι ε, το, ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων. Έχουν υποβληθεί και εδώ πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες ζητούν δραστική μείωση της περίοδου κράτησης διατήρησης των στοιχείων. Έχουμε προτείνει εμείς μια συνολική περίοδο διατήρησης στοιχείων πενταετή. Κάποιες από τις τροπολογίες ε, ζητούν ε, τρεις, δεκατρεις μέρες ε, ή τρεις μήνες. Το είπαμε και στο παρελθόν και θα το επαναλάβω και σήμερα ότι δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος αξιολόγησης του, της σωστής ορθής περίοδου διατήρησης των στοιχείων. Εμείς επιλέξαμε την πενταετή περίοδο διότι ε, η εμπειρία των αστυνομικών αρχών ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πενταετής είναι και η περίοδος επιβίωσης των ε, εγκληματικών ομάδων. Ποικίλουν λοιπόν οι προτάσει. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι 3, οι 13 μέρες και οι πέντε μήνες σαφώς δεν είναι επαρκής περίοδος. Όσον αφορά τις εσωτερικές πτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο κύριος Κυρκόπ στο θέμα αυτό. Στην πρότασή μα δεν έχουμε περιλάβει ε, τις ε, εσωτερικές πτήσεις. Η πρότασή μας περιορίζεται στις διεθνείς πτήσεις. Όμως αναγνωρίζομαι ότι ε, η προστιθέμενη αξία της ασφάλειας των εσωτερικών πτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική και επομένως θα αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο ε, να συμπεριλάβουμε και τις εσωτερικές πτήσεις σε δύο χρόνια μετά την ε, θέση σε ισχύ ε, της, του συστήματος PNR για τις διεθνείς πτήσεις. Οι εσωτερικές πτήσεις αφορούν τα δύο τρίτα των πτήσεων, επομένως είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πτήσεων είναι επικίνδυνο να συμπεριληφθούν και εσωτερικές πτήσει από την αρχή γιατί το σύστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, βαρύ, δύσκολο στην εφαρμογή του και επομένως θεωρούμε ότι η καταβήμα προσέγγιση είναι καλύτερη η προσέγγιση που εμφανίζεται σε κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες στοχεύουν ακριβώς στην ρητή, στο ρητό αποκλεισμό, στη ρητή εξαίρεση των ε, εσωτερικών πτήσεων ε, αποκλείοντας την ενδεχόμενη συμπερίληψη των πτήσεων αυτών στην αναθεώρηση που θα γίνει μετά από δύο χρόνια όπως είπα προηγουμένως θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή η τοποθέτηση το μόνο που είπαμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση αργότερα και εάν και εφόσον αποφασιστεί να συμπεριληφθούν οι πτήσεις αυτές, τότε θα υπάρξει μια νέα πρόταση από της οποίας θα έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε. Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε, αλλά το να αποφασίσουμε από τώρα να αποκλείσουμε ολοκληρωτικά τις εσωτερικές πτήσεις θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ε, ρίζοσπαστικό και δεν το δεχόμαστε. Αυτά είχα να πω μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν από την Προεδρία, μήπως θα ήθελε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο σημείωσε τις πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Όπως ξέρουμε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν συμφωνούν κατά ανάγκη σε όλα τα θέματα που θίγουν και οι τροπολογίες. Το Συμβούλιο ανισχύει ιδιαίτερα διότι κάποιες από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν θα περιορίσουν δραστικά το εύρος και την ε, λειτουργική χρήση των πληροφοριών του συστήματος. Ήδη αναφέρθηκε και από τον κύριο το θέμα του περιορισμού της χρήσης του PNR μόνο για αδικήματα τρομοκρατίας και όχι για την πρόληψη και ανείχνευση και διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων όπως και η Επιτροπή και ο εισηγητής. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα χάσουμε ε, μια σημαντική προστιθέμενη αξία του συστήματος. Επίσης, ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν με τον εισηγητή ότι ε, οι ενδοενωσιακές πτήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής και βεβαίως η ενεργή χρήση του συστήματος. Η Επιτροπή έδωσε μια ε, σειρά από εξηγήσει γιατί πρέπει να, είμαστε, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίε, να χρησιμοποιούμε με τον πιο ενεργό τρόπο τα στοιχεία αυτά. Αλλά φυσικά υπό αυστηρέ προποθέσει. Το λαμβάνει ιδιαίτερα και αυτό το Συμβούλιο υπόψη. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω στις ε, μελλοντικές διαπραγματεύσεις μας, αλλά έχει κάθε εμπιστοσύνη το Συμβούλιο, λόγω της πολιετούς πείρας μας αντιμετώπισης του θέματος αυτού, ότι θα διεξαγάγουμε επικοδομητικό διάλογο για το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, Το θέμα θα υποβληθεί στο Συμβούλιο αύριο για μια πρώτη γενική συζήτηση και κατόπιν ελπίζουμε να έχουμε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις και με το Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα να λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές που το ζήτησαν. Η κυρία Σούμε Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν πολύ σημαντικές τροπολογίες. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ότι υπάρχει ανησυχία σε όλες τις πολιτικές ομάδες για την πρόταση αυτή. Έχει να κάνει με την περίοδο χρήση των στοιχείων, αποθήκευση των στοιχείων, το πεδίο εφαρμογής, πώς θα γίνεται η συλλογή των στοιχείων, αλλά στην ουσία αυτό που τίθεται εν αμφιβόλο είναι η φιλοσοφία πρόληψης των αδικημάτων. Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα της ε, πρότασης αυτής. Έτσι ακριβώς το υπογράμμισε και ο Ευρωπαίος ε, Επιτηρητής Προστασίας των Δεδομένων που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και έκανε μια πολύ αρνητική έκθεση για αυτήν την πρόταση. Και αυτό είπε και η ομάδα εργασίας για το άρθρο 29 της παλιάς οδηγίας προστασίας των δεδομένων. Η ομάδα αυτή εργασίας δεν, ήταν μόνο, δεν, δεν αποτελεί το μόνο από νομομαθείς, αλλά και από τους διευθυντές των 27 υπηρεσιών προστασίας δεδομένων των χωρών μας. Όταν λοιπόν ε, αμφισβητεί και η ομάδα αυτή και ο Ευρωπαίος επιτηρητής, ε, πρέπει να υπάρχουν λόγοι. Ας εξετάσουμε την ε, απαρχή της ε, αρχής της ε, αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Αυτές είναι οι αρχές που έχουν στόχο να καταργήσει τη βαρβαρότητα των παλιών ποινικών κωδίκων, των προδημοκρατικών καθεστώτων. Να ξανακάνουμε τώρα πάλι τέτοια ανάλυση για ένα σημερινό νομοθέτημα το είπα επανειλημμένα. Θα έπρεπε να γυρίσουμε στο ρωμαϊκό δίκαιο. Γιατί εκεί γεννήθηκαν αυτές οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Α, είναι εδώ ο κύριος Κέρκο. Θα μπορούσα να αναφερθώ στον ε, μεγάλο Βρετανό Ρόμπερτ Πιλ που αναφέρθηκε τις αρχές αυτές. Ίσως θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο Μοντεσκέ, όταν έλεγε ότι κάθε νόμος που δεν προκύπτει από αναγκαιότητα είναι τυραννικός. Μπορεί λοιπόν να προκύψει κίνδυνος ότι η προσπάθεια πρόληψης ενός εγκλήματος για την οποία δεν υπάρχει αναγκαιότητα γεννά τυραννία. Αυτή είναι πράση του Τσέζαρε Μπεκαρία. Καλύτερα λοιπόν, έλεγε ο Μπεκαρία, να είναι ένας ένοχος ελεύθερος, προτιμότερο αυτό, παρά να είναι ένας αθώος φυλακή. Γιατί ξέρετε τις ε, συνήθειες που εγκαταλείψαμε με τους νέους ποινικού κώδικες, τις κακές ειδικές κράτησης, τους βασανισμούς κτλ. Όπως έλεγε λοιπόν ο Μπεκαρία, η πρόληψη ενός αδικήματος πρέπει να βασιστεί πάνω στην ασφάλεια και τη σιγουριά και όχι την σοβαρότητα των τιμών. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις, χρειαζόμαστε αποδείξεις. Γι' αυτό μιλάμε για τις αρχές δικαίου που υπάρχουν για να μην θεωρούνται όλοι οι πολίτες ύποπτοι. Αυτή είναι η βαρβαρότης που δημιουργείται με βάση κάποιες προσπάθειες που γίνονται για την πρόληψη του εγκλήματος. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Όλοι οι πολίτες θεωρούνται ύποπτοι. Αυτή η διαμάχη που υπάρχει για το θάνατο του Τρέβορ Μάρτιν, αυτού του νέου 17 ετών που επειδή φοράει κουκούλα και επειδή κουνιόταν ακούγοντα μουσική, θεωρήθηκε ύποπτο και τον ε, δολοφόνησε κάποιο από μια ομάδα πολιτοφυλάκων ιδιωτικών. Δεν μπορεί να είναι αυτή η κοινωνία μα. Οι πολίτε μα ταξιδεύουν. Επειδή ταξιδεύουν δεν είναι ύποπτοι. Επειδή μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο. Η φιλοσοφία λοιπόν για την πρόληψη ενός αδικήματος πρέπει να είναι η σωστή για να υπάρχει πρόληψη που να είναι αποτελεσματική, που να βασίζεται στην νομική ασφάλεια και στη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Αυτό που κάνουμε είναι παρόμοιο με το αμερικανικό PNR και τις συμφωνίες που κάναμε με τους Αμερικανούς και θέτουμε κινδύνο τι αξίε που έχουμε περασπιστεί στην Ευρώπη και που δυστυχώς ε, δεν τη συμμερίζονται οι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί έχουν αυτή την αρχή της ε, επιβολής της ποινή του θανάτου, θεωρούν ύποπτους όλους τους πολίτες τους μια σειρά από νομοθετήματα και απόψεις που εμείς τους δικούς μας ποινικού κώδικες δεν τους διατηρούμε. Υπάρχει η τρομοκρατία βεβαίως. Και βεβαίως Πρέπει να υπάρχουν κάποια έκτακτα μέτρα γι' αυτό, γιατί βεβαίω πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ε, ταξιδιωτών και πρέπει να λάβουμε λοιπόν εξαιρετικά ειδικά μέτρα και οι ποινικοί κώδικες των χωρών όπου υπήρξαν φαινόμενα τρομοκρατία συμπεριλαμβάνουν και τέτοια μέτρα. Για παράδειγμα, η χρήση των μετανοούντων, για παράδειγμα, οι υποκλοπέ τηλεφωνικών επικοινωνιών. Υπάρχουν. Αλλά αυτά τα μέτρα είναι επειδή υπάρχει άμεσο κίνδυνο και για να μπορέσουμε να συλλάβουμε επαυτοφόρο τους εγκληματίες. Αυτή πρέπει να είναι η βάση της εξαιρετικότητας των μέτρων. Θα πρέπει να υπάρχει και σαφής παρέμβαση της δικαιοσύνης. Μόνο ένας δικαστής μπορεί να ξεκινήσει την εφαρμογή αυτών των εξαιρετικών μέτρων και να ενημερώνεται πάντα ο δικαστής όταν χρειάστηκαν να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την παρέμβασή του. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Πρέπει, δεν θα πρέπει να είναι κυβερνητικές οι αρχές που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, πρέπει να εμπλέκονται οι δικαστικές αρχές, όπως λέγεται σε κάποιες τροπολογίες, πρέπει να γίνει μια δικαστική έρευνα που να επιτρέπει μετά τη συλλογή στοιχείων, Ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορεί να γίνει συλλογή στοιχείων όταν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της εξαιρετικότητας. Είναι λοιπόν πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ναι, ναι, κατά λίγο, κατά λίγο, Γιατί δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανένα άλλο, λέει ο πρόεδρο. Κοιτάξτε, υπάρχουν 500 τροπολογίε, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αλλά όταν μιλάει για νομιμότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για νομιμότητα, η νομιμότητα αποτελείται από του νόμου. Πηγή νομιμότητα δεν είναι το, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και αν είναι αρμόδιες για το θέμα αυτό, δεν είναι πηγή νομιμότητας. Και είναι πολύ ε, αξιοσημείωτο ότι η συζήτηση για την προστασία των δεδομένων θα έρθει μετά από αυτό το πακέτο για το PNR. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, λυπάμαι πραγματικά, αλλά θα φύγει ο εισηγητής. Άρα πρέπει να μπορέσουν ε, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Φόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πολύ μεγάλος αριθμός τροπολογιών καθιστά σαφές ότι όλοι δεν ξέρουμε πού πάει αυτό το ταξίδι με αυτό το νομοθέτημα από το συγκεντρωτικό μοντέλο στο αποκεντρωμένο μοντέλο και στην ομάδα μου δεν έχει διαμορφωθεί άποψη. Διότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Είναι δυσνόητα τα κείμενα αυτά. Νομίζω ότι ο εισηγητής έκανε μια θαυμάσια έκθεση. Υπάρχει προστιθέμενη αξία από ό,τι μπορώ να καταλάβω μέχρι τώρα. Στην ανάλυση των στοιχείων PNR Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε ιδιαίτερα, να... δεν πρέπει όλα να τα αναλύουμε, αλλά να μην περιορίσουμε ό,τι μπορεί να αναλυθεί και να γίνει αντικείμενο επεξεργασία. Και γι' αυτό με τι τροπολογίε μου επιχείρησα να προσθέσω αξία και σε ένα κεντρικό στοιχείο του συστήματος. Είναι απόλυτα αναγκαίο, επιγόντω αναγκαίο, εφόσον ε, περνάμε από 27 κράτη-μέλη σε ένα κεντρικό σύστημα, Πρέπει να υπάρξει αυτή η διόρθωση. Δεν ξέρω πόσο γίνεται ευρέως αποδεκτή αυτή η ιδέα, αλλά κανείς δεν μου ανέφερε κανένα επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ότι θα είναι δύσκολο βεβαίως, ότι θα υπάρξουν δυσχέρειες προσαρμογής βεβαίως. Αλλά κανείς δεν μου είπε ότι θα ήταν αδύνατο. Συνολικά για την κατάσταση, επειδή το θέμα αυτό είναι συνολικά επίμαχο, να επιχειρήσουμε να βρούμε μια ελάχιστη κοινή βάση. Ίσως η δημιουργία ενός PNR εθελοντικά ε, τα κράτη-μέλη, ίσως θα μπορούσε να είναι αυτή η βάση, θα μπορούσε να ισχύσει έτσι λοιπόν εθελοντικά και για τις ενδοενωσιακές πτήσεις. Αλλά όταν δημιουργηθεί τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, βασίζεται σε ορισμένα κριτήρια που να ισχύουν για όλους. Δύσκολο ξέρω ότι είναι ότι για τις αεροπορικές εταιρείες θα είναι δύσκολο να αποφασίζουν τι στοιχεία να στείλουν και σε ποιον. Επιπλέον, αν ε, υιοθετήσουμε ένα τέτοιο εθελούσιο σύστημα, η δικτύωση θα ήταν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την επιτυχία του. Να αρκεστώ σε αυτά, αλλά συνολικά παρακαλώ, εφόσον έχουμε τις τροπολογίες, να κάνουμε μια προσπάθεια να οδεύσουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί προς το παρόν αποκλίνουν πολύ οι κατευθύνσεις μας. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είναι θέμα που αφορά την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλβαρο. Ευχαριστώ. Η υποβολή τόσων πολλών τροπολογιών οφείλεται ότι στην ομάδα μου Οφείλεται λοιπόν στο ότι είμαστε θεμελιωδώς κατά αυτής της πρότασης, απορρίπτουμε κάθε τμήμα της. Νομίζω ότι είναι σαφές. Με συγχωρείτε και συνάδελφοι των υπηρεσιών που χρειάστηκε να ασχοληθείτε με τόσες πολλές τροπολογίες. Όμως, από αυτά που ακούσαμε ενισχύεται η άποψή μας. να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή σε όλου του τομεί ε, τρομοκρατία και οργανωμένου κλίματος, ε, διερωτώμε. Ξέχουμε ήδη βάση δεδομένων για τι ε, προξενικές θεωρήσεις. Εάν επιτρέψουμε τα κράτη-μέλη, ε, τα οι τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση, αποφασίσαμε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα θεωρώντας ότι και εμείς θα ωφεληθούμε, θα λάβουμε πληροφόρηση. Καλό είναι να δούμε τα στοιχεία τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε καλή και πολιτισμένη και επιτυχημένη αστυνομική συνεργασία. Έχουμε τη συμφωνία του ΠΡΙΜ, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, έχουμε φτιάξει τη Europol, είναι, μια, είναι ένας οργανισμός που έχει ευρύ ε, πεδίο λειτουργίας, έχουμε συνεργασία των μεθοριακών αρχών. Πού είναι λοιπόν η προστιθέμενη αξία. Έχουμε τόσα όργανα. Γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια συμφωνία. Όλες οι συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες όπως είπα και το SWIFT και με τις ΗΠΑ βασίστηκαν στο ότι θα ωφεληθούμε κι εμείς. Είναι καλύτερο λοιπόν ε, αυτή η αμοιβαιότητα να επεκταθεί περαιτέρω. Ούτω ώστε να έχουμε δυνατότητα έτσι να αποκτήσουμε τα στοιχεία. Κοιτάξτε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί τότε οι τρομοκράτες να μην πάρουν το τρένο, όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Τότε μετά μπορεί να πούνε ωραία, να δούμε και με τους ε, ταξιδιώτες το τρένο. Γιατί κάποιο μπορεί να πάει από τη Βαρσοβία στο Βερολίνο, τότε και αυτό θα πρέπει να αποσταλούν τα στοιχεία του. Θα έχουμε μετά PNR και για τα τρένα. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν, δεν νομίζω ότι, ότι έχει σπουδαία έννοια. και για πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούνται τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κανένας μαθηματικός τύπος. Ε, ο καθένας λέει κάτι, τρει, έξι, εννιά μήνες. Αλλά υπάρχει ένας πολύ απλός ε, τρόπος να καταλάβουμε τι προθεσμία. Η χρήση. Οι περισσότερες αρχές μπορούν να μας πούνε για πόσο χρόνο θεωρούν ότι είναι χρήσιμα τα στοιχεία. Εγώ από ό,τι άκουσα διάφοροι ε, εισαγγελεί μου είπαν ότι τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα τρει με έξι μήνες. Αυτοί ξέρουν από την εμπειρία του πόσο καιρό είναι χρήσιμα τα στοιχεία αυτά. Με βάση λοιπόν την εμπειρία των, των ειδικών θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε το σωστό στοιχείο. Κάτι νόμου τους άλλους δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί η πρότασή μου τους άλλους δεν η, συγγνώμη, η ομάδα μου δεν πρόκειται να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη η εξέβρεση ε, συμβαστικών λύσεων. κύριος Άλμπεχτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ως πράσινοι και εμείς έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες και εμείς θεωρούμε την πρόταση όσο έχει τώρα από την Κομισιόν και όπως συζητείται στο Συμβούλιο με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα τη θεωρούμε απαράδεκτη με εξέπληξε κάπως ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε βασικά συνταγματικά θέματα και προστασία δεδομένων, αγνοώντας τα. Φυσικά μπορούμε να πούμε στην πρόταση αυτή, όπου γίνεται επέκταση του πεδίου εφαρμογής, μιλάμε για ενδονοσιακές πτήσεις κτλ. Όλα αυτά τίθενται ως πρόληψη. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι η πρόταση αυτή οπωσδήποτε θα ακυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα Εθνικά Δικαστήρια. Δεν είναι δυνατόν εμείς αρχές που λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις ως Συμβούλιο Υπουργών. Δεν καταλαβαίνω πόσο μικρή ευαισθησία έχει το Συμβούλιο των Υπουργών για το θέμα αυτό. Και εμεί εδώ ω βουλευτέ δεν καταλαβαίνω γιατί πολλοί έχουμε τόσο μικρή ευαισθησία για την νομική βάση και για τα συνταγματικά μα όρια. Και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Θα πρέπει να κάνουμε μια πιο θεμελιώδη και φιλοσοφική συζήτηση για το θέμα αυτό για να καταλάβουμε τι είδου μέτρα είναι αυτά. Είναι μέτρα που πολύ πριν διαπραχθεί ένα αδίκημα αρχίζουν να λειτουργούν αφορούν όλους τους πολίτες τα στοιχεία των πολιτών θα είναι για πέντε χρόνια προτείνεται τα στοιχεία για οποιαδήποτε πτήση που θα έχουν κάνει αγαπητοί συνάδελφοι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα ξέρετε ότι η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των δεδομένων έχει προβλήματα από το συνταγματικό δικαστήριο η γερμανική κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες ή μόνατες δεν θα μπορέσει να υποβάλει νέο νόμο διότι τα όρια, τα συνταγματικά όρια για την άσκοπη συλλογή και αποθήκευση στοιχείων είναι τόσο ψηλά στις προτάσεις που είναι απαράδεκτα. Μιλάμε τώρα για αποθήκευση στοιχείων για έξι μήνες και για επεξεργασία των στοιχείων από ιδιωτικές εταιρείες για να αξιοποιούνται μετά από την έγκριση του δικαστή, όπως είναι αυτή η πρόταση. Τώρα λέγεται ότι μια κρατική αρχή για πέντε χρόνια. αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια οποιασδήποτε συνταγματικής συζήτησης, οποιασδήποτε συζήτησης για την προστασία των δεδομένων. Παρακαλώ, με βάση τις πολλές τροπολογίες που έχουν υπάρξει, να ξανασυζητήσουμε για την έννοια, την αναγκαιότητα τέτοιων ευρωπαϊκών μέτρων και να μην συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοθέτημα. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί τι ρόλο παίζει. Να πούμε τι κάνουμε έναντι των πολιτών της Ευρώπης. Τους αντιμετωπίζουμε με θεμελιώδη δυσπιστία. Όλους, εάν εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Και αν θέλουμε και τις εσωτερικές πτήσεις της Ένωσης να τις συμπεριλάβουμε θεμελιώδη δυσπιστία έναντι των πολιτών μας. Τους θεωρούμε υπόπτους, όλους, χωρίς αίτιο. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχει σχέση η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα, δεν θα δώσει καμία προστιθέμενη αξία. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που να αιτιολογεί τέτοια μέτρα. Ποια είναι η αναγκαιότητα, ποια είναι η αναλογικότητα. Δεν τα βλέπω. Είναι σκανδαλώδες να επεκτείνεται τόσο πολύ το πεδίο εφαρμογής, να συμπεριλαμβάνεται η σοβαρή εγκληματικότητα ως συμπροματικό πρόσθετο θέμα, να σκεφτούμε σε τι βαθμό θα το συμπεριλάβουμε. Δείτε πόσο δύσκολο είναι να καθορίσουμε την σοβαρή κλιματικότητα και τα όρια της. Βεβαίω υπάρχει κίνδυνο από τον χαρακτηρισμό, αυτό το profiling. Έχουμε προβλήματα με την αποθήκευση. Γιατί για όνομα του Θεού πέντε χρόνια. Κανεί δεν μα το εξήγησε. Εσεί είπατε όχι τρει μέρε, όχι τρει μήνε. Αλλά γιατί πέντε χρόνια σα ρωτάω. Για όνομα του Θεού. Γιατί πέντε χρόνια. Να μην μιλήσω τώρα για τρίτες χώρες, για την ασφάλεια των δεδομένων και πολλά άλλα που ρυθμίζονται με πολύ προβληματικό τρόπο και στην πρόταση της Κομισιόν και στην έκθεση τη δική μας. Πρέπει να πω Έχω υποβάλει την τροπολογία 38, όπου η ομάδα μας λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση, αν μείνει έχει. Για μας δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει βάση για συμβιβασμού. Είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται. Το καλύτερο θα ήταν η Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της. Σας κατευχαριστώ. Έχουν τεθεί θεμελιώδη ερωτήματα εδώ μέσα. Η κυρία Σίπα. Ευχαριστώ να περιοριστώ σε δύο-τρία σημεία γιατί πολλά ήδη αναφέρθηκαν. Όλοι θέλουμε να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας με αναλογικότητα. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι αν όντως αξιοποιείται, αν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε κάθε μέσο για κάθε στόχο. Θυμηθείτε συνάδελφοι, γιατί ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση την ξεκινήσαμε για να, να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα συστήματα SWIFT και τα λοιπά και PNR στι ΗΠΑ για την τρομοκρατία. Τώρα μιλάμε για την τρομοκρατία, για σοβαρό οργανωμένο διαμεθοριακό έγκλημα και ακόμη για σοβαρή εγκληματικότητα ή γενικά για εγκληματικότητα. Και δεν είναι μόνο πρόβλημα για τις αεροπορικές εταιρείες και για την αποθήκευση, και για τις αστυνομικές αρχές, τα στοιχεία αυτά θα τα αξιοποιούσαν για ό,τι να είναι. Αυτό το τόσο ευρύ ε, πεδίο εφαρμογή είναι σίγουρα υπερβολικό. Και επίσης, προς τα πού αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας. Το PNR είπαμε ότι αφορά τις ε, διεθνείς πτήσεις, ε, τώρα μιλάμε για εσωτερικές πτήσεις της Ένωσης, τώρα μιλάμε για ορισμένους, για τους επιβάτες καράβια, για τρένα. Γιατί να μην ε, μπαίνουμε και σε κάθε αυτοκίνητο για να πάρουμε τα στοιχεία του οδηγού. Πολλοί είπανε κοστίζει πολλά, γι' αυτό θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος, τότε γιατί να μην περιορίσουμε το, το, πεδίο εφαρμογής. Ξεκινήσαμε με τρομοκρατία και την οργανωμένη εγκληματικότητα και αν δούμε ότι ε, αποδίδει το σύστημα τότε να το επεκτείνουμε. Αν δούμε πώς θα εφοδιάσουμε οικονομικά και με προσωπικό τις υπηρεσίες αυτής, τις υπηρεσίες αυτές, αναρωτιέμαι με βάση και τις υπάρχουσες αστυνομικές και άλλες αρχές συνεργασίας, εάν χρειάζεται να δαπανίσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την εγκληματικότητα τελευταίο. Προστασία των δεδομένων. Εάν υπάρξει μια τέτοια οδηγία, πρέπει οπωσδήποτε η νομική βάση να διευρυνθεί. Να συμπεριλάβει το άρθρο 16, προστασία των δεδομένων. Και να αναφέρω το πρόγραμμα εφαρμογής της πρωτοβολίας της Στοκχόλμης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς περιορισμούς, να είναι συγκεκριμένα και αποτελεσματικά η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας είναι πολύ σημαντική. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την προστασία τους ακόμη και για τον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης εγκληματικότητας. Και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες στον τομέα αυτό. Όχι να διασφαλίσουμε, να ενισχύσουμε. Και δεν είναι μόνο θέμα ε, προθεσμίας αποθήκευσης, αλλά και αναλογικότητα της χρήσης των στοιχείων. Ευχαριστώ κύριο Ζαγκάρ. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω σε δύο θέματα που είχαν τεθεί στην προηγούμενη συζήτησή μας του θέματος. Γιατί τα άλλα τα είπαν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τι είδους εγκλήματα θέλουμε να παρακολουθούμε. Αν δεχόμασταν την έννοια μίας ελάχιστης φυλάκισης τριετούς, τότε θα μιλούσαμε για πλημελήματα, όχι για εγκλήματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω και εξακολουθώ γιατί θέλουμε να ελέγξουμε ή να παρακολουθήσουμε τον διεθνή εγκληματία που έκλεψε ένα ποδήλατο στο Αάχεν τη στιγμή επειδή λέει είχε εκφράσει την πρόθεσή του αυτή στις Βρυξέλλες. Μα προθέσεις παρακολουθούμε εδώ. Τα εγκλήματα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε είναι τόσο σοβαρά ώστε ήδη έχουν σοβαρότερες κυρώσεις. Δεν χρειάζεται εδώ να προβλέψουμε και τι κυρώσεις και τι φυλάκιση. Μετά κατά πόσον όλα αυτά θα εφαρμοστούν και στις εσωτερικές πτήσεις. Εγώ είμαι κατά της ιδέας αυτής αλλά συνδέεται με κάτι άλλο που θέλω να το απαντήσει το Συμβούλιο ίσως και η Επιτροπή ή μάλλον η Επιτροπή επιτροπη ίσως και το Συμβούλιο ε? δηλαδή τις ε, πτήσεις χαμηλού κόστους τις φτηνές πτήσεις οι οποίες λένε ότι δεν θα καλύπτονται ούτως ή άλλως γιατί αυτές έχουν δικό τους σύστημα PNR Μερικές από αυτές τις φτηνές εταιρείε πετούν και μέσα και έξω από την Ένωση και άρα αν τυχόν παρελπίδα καλύπταμε και τις εσωτερικές πτήσεις τότε θα έπρεπε να εξετάσουμε και κατά πόσον θα καλύψουμε τις φθηνές αεροπορικές εταιρείες, διότι εάν όχι, τότε και οι πραγματικά διεθνείς πτήσεις και οι εσωτερικές θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σύγχυσης. Ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε ο εισηγητής, τον χάσαμε. Και γι' αυτό ίσως η Κομισιό να μας απαντήσει. Η κυρία Βασιλιάδου. Σημειώνω όλα αυτά που ακούστηκαν και θα απαντήσω μόνο στο τελευταίο ερώτημα του κυρίου Έγγελ για τις χαμηλού κόστους εταιρείες οι οποίες θα καλύπτονται. Δεν έχει σημασία αν έχουν δικό τους PNR. Ο δικός μας ορισμός του τι είναι PNR θα καλύπτει και αυτές. Επομένω θα συμπεριλαμβάνονται και αυτές. Ευχαριστώ για τη συζήτηση την οποία σημειώνουμε δεόντως. Α, σας ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλιά σας. Κυρία Όκεν, παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Δεν θα επισελθώ σε μεγάλες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω απλώς ότι το θέμα θα υποβληθεί αύριο στο Συμβούλιο το οποίο θα εκφραστεί συγκεκριμένα για το θέμα των εσωτερικών πτήσεων και για την περίοδο διτήρηση των στοιχείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και τον τριμερή διάλογο. Τώρα τελείωσε η πρωινή μας συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στα 3 με τον Έλληνα Υπουργό.